Καλημέρα σε όλους. Ξεκινάει η συνεδρίαση της Ολομέλειας. Θα ξεκινήσουμε με τα συμπεράσματα και τη, το, τη συζητάσεις της σκέψεως των διακοινοβουλευτικών επιτροπών. Ε, θα διαρκέσει περίπου μισή ώρα. Μετά θα έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε τον Έλληνα Υπουργό των Οικονομικών, τον Γιάννη Στουρνάρο, ο οποίος βέβαια είναι και πρόεδρος του ΕΚΟΦΗΝ. Θα ακολουθήσει η ανταλλαγή απόψεων και το κλείσιμο θα γίνει με την ομιλία του κυρίου Κάρας και τη δική μου που θα κλείσω και τη συνδιάσκεψη. Θα ήθελα να σας παρακαλέσω να ξεκινήσουμε όπως και στις προηγούμενες συνεδριάσεις μας επειδή θα υπάρξει κατάλογος ομιλητών να έχουμε τέσσερις ομιλητάς από τα Εθνικά Κοινοβούλια και έναν ομιλητή από, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Yes. okay. Ναι, ναι, όχι, ε, αυτό είναι και τη Οκ, ποιος είναι το Η κυρία Σάρον Μπόλ παίρνει το λόγο. Ε, yes. Οκ, okay, το λόγο έχει η κυρία Σάρον Μπόλς για 10 λεπτά. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Μόλις ολοκληρώσαμε και εμείς όπως και οι υπόλοιπες κοινοβουλευτικές επιτροπές τη συζήτηση που κάναμε για δύο συγκεκριμένα ζητήματα, αποτελεσματικό σύστημα φόρου θέμενη αξία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Καταλαβαίνετε ότι αποτελεί ένα πολύ σημαντικό πόρο εισοδήματο για την Ευρωπαϊκή Ένωση το ζήτημα αυτό και μολονότι έχουμε πετύχει πολύ σημαντικέ επιτυχίε όσον αφορά το παγκόσμιο σύστημα φόρου θέμενη αξία και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αναγνωρίζουμε όλοι ότι υπάρχουν ακόμα πολύ μεγάλε αδυναμίε, καθώ επίση και ένα υψηλό βαθμό πολυπλοκότητο. Πρέπει λοιπόν το σύστημα αυτό το νέο εφαρμόζεται πολύ απλά η συνταγή φαίνεται να αναπλεί, να καταργηθούν ουσιαστικά εξαιρέσει, να καταφέρουμε να κάνουμε το σύστημα πιο αποτελεσματικό και πιο συνεκτικό. Ωστόσο όμως όταν βλέπουμε τους υφιστάμενους συντελεστές, καθώς επίσης και τους μηδενικούς συντελεστές που υπάρχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς επίσης και όλες αυτές τις εξαιρέσεις, συνειδητοποιούμε ότι υπάρχει ένα τεράστιο διοικητικό άχθος στα πλαίσια του συστήματος αυτού, τόσο για τις εθνικές εφορίες όσο και για τις επιχειρήσεις, τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θεωρούμε βέβαια ότι με τις προτινόμενες από εμά αλλαγές υπάρχουν διάφορα προβλήματα σε διάφορα κράτη-μέλη τα οποία προσπαθούν να προτάξουν διάφορες ε, εθνικές ενστάσεις, οι οποίες πολλές φορές έρχονται ακόμα και από βουλευτές. Πράγμα το οποίο καθιστά δύσκολο το έργο μας και για αυτό το λόγο έχουμε ένα κενό 250 εκατομμυρίων ευρώ όσον αφορά τον φόρο προστιθέμενης αξίας και υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό το οποίο έχει να κάνει με την απάτη στο φόρο προστιθέμενης αξίας. Ο φόρος προστιθέμενης αξίας ενδεχομένως να μην λειτουργεί πολλές φορές διασυνοριακά για πολλές εταιρείες ή μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Γενικότερα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υποστηρίζει την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο στρατηγικό της έγγραφο και συμφωνεί με τον μηχανισμό έγκαιρη προειδοποίηση και ανάληψη δράση όσον αφορά την απάτη για το φόρο προσθέμενη αξία, καθώ επίση και με του νέου κανόνε που θα πρέπει να αρχίσουν να ισχύουν από το 2015 και μετά. Θεωρούμε ότι θα πρέπει να υπάρχει ένα συγκεκριμένο ποσοστό επιστροφή του φόρου προστιθέμενη αξία σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ακριβώ αυτό επεξεργαζόμαστε στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και θεωρούμε να, θέλουμε να έχουμε παντού στην Ευρωπαϊκή Ένωση κοινέ κατευθυντήριε γραμμέ. Προσπαθούμε επίση να δούμε πώ εξελιχθούν τα πράγματα στο μέλλον, στα πλαίσια τη Επιτροπή μα. Στι συζητήσει τώρα που κάναμε, επικεντρωθήκαμε κυρίω στο ότι χρειάζεται περισσότερο χρόνο για την υποβολή εκθέσεων, καλύτερη ανταλλαγή στοιχείων και δεδομένων άμεσα στα κράτη-μέλη όσον αφορά το φόρο προστιθέμενη αξία πάντα. Ελπίζουμε ότι θα καταφέρουμε να πετύχουμε το απαραίτητο κατόφλι ανταλλαγή πληροφοριών. Υπάρχουν συγκεκριμένοι μορφότυποι που χρησιμοποιούνται από ορισμένα κράτη-μέλη όσον αφορά την επιστροφή του φόρου θέμενη αξία. το γεγονός ότι ο μορφότυπο αυτός δεν είναι κοινό για όλα τα κράτη-μέλη δημιουργεί ακόμα διάφορα προβλήματα, Νομίζω ότι ε, θα πρέπει να έχουμε έναν κοινό τρόπο ανταλλαγής ε, πληροφοριών προκειμένου να καταφέρουμε να εξασφαλίσουμε την απόδοση του φόρου προσθέμενης αξίας παντού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πιστεύω ότι μέσω της πιο αποτελεσματικής ανταλλαγής πληροφοριών θα είμαστε σαφώς σε μια καλύτερη θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα γίνουμε πολύ πιο αποτελεσματικοί και νομίζω ότι θα ήταν θετικό να είχαμε και μία ομάδα εργασίας η οποία θα μπορούσε να ασχοληθεί ακριβώς με τα ζητήματα αυτά θα ήταν πολύ θετικό να είχαμε μια τέτοια ομάδα εργασία στην επόμενη κοινοβουλευτική θητεία και να καταφέρουμε να έχουμε επίση περισσότερε συνεδριάσεις μέσω τηλεδιάσκεψη ενδεχομένω και με πολλά κράτη-μέλη στα πλαίσια της επόμενης κοινοβουλευτικής θητείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Κατά αυτόν τον τρόπο θα είμαστε σε συνεχή επαφή με τα κράτη-μέλη αλλά και με τα εθνικά κοινοβούλια. Είπαμε επίσης ότι θα πρέπει να υπάρχει μια ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών όσον αφορά τις ε, διαφορετικές αλλαγές πρέπει να γίνουν στα κράτη-μέλη. Στα πλαίσια της ε, ετήσιας επισκόπησης ανάλυσης Ευρωπαϊκής Επιτροπής είδαμε ότι υπάρχουν συγκεκριμένα μέτρα τα οποία θα μπορούσαν να εφαρμοστούν προκειμένου να γίνουν οι εθνικές διοικήσεις πολύ πιο αποτελεσματικές. Καλούνται πολλά κράτη-μέλη να εφαρμόσουν διαφορετικέ μεταρρυθμίσεις και να καταφέρουν να εξηγιάνουν στα πλαίσια του νέου κύκλου Ευρωπαϊκού, Ευρωπαϊκού τα δημόσια οικονομικά του. Οι μεταρρυθμίσει αυτέ είναι απαραίτητε προκειμένου τα οικονομικά των κρατών μελών να γίνουν βιώσιμα. Αν δεν γίνουν όμω οι μεταρρυθμίσει αυτέ, αυτές, τότε ενδεχομένω να οδηγηθούμε σε νέα ανάληψη κινδύνου από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα από το μηχανισμό ESM. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να βρούμε την κατάλληλη ισορροπία για τις μεταρρυθμίσεις που θα πρέπει να γίνουν και θα πρέπει οι μεταρρυθμίσεις που θα έχουν ως στόχο την οικονομική ανάπτυξη να προωθούν επίσης τη δημοσιονομική εξυγίανση, ενώ θα πρέπει να υπάρχει ένας καλύτερος μακροοικονομικός καταμερισμός των μεταρρυθμίσεων αυτών. Προσπαθήσαμε να έχουμε μια συμμετρική προσέγγιση όσον αφορά την μακροοικονομική προσαρμογή και είπαμε επίσης κατά τη διάρκεια των συζητήσεών μας ότι οποιοδήποτε πιστωτής, είτε μιλάμε για τράπεζες, είτε για άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, είναι πάρα πολύ σημαντικό να θέτει τις απαραίτητες προϋποθέσεις προκειμένου να διασφαλίσει ότι θα καταφέρει να επανακτήσει τα χρήματα τα οποία δανείζει. Ορισμένα κράτη-μέλη αυτή τη στιγμή καταβάλουν πολύ σημαντικές προσπάθειες προκειμένου να καταφέρουν να εφαρμόσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα μέτρα αυτά μακροπρόθεσμα θέλουμε τα ζητήματα αυτά να μπορούν να διευθετούνται στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποκλειστικά, χωρίς να χρειάζεται η παρεμβολή εξωτερικών διεθνών οργανισμών. Άλλα ζητήματα τα οποία θίξαμε ήταν το ότι θα πρέπει να δημιουργηθούν τα απαραίτητα κίνητρα και μηχανισμοί αποζημίωσης αντιστάθμισης όσον αφορά την εφαρμογή των διαφορετικών μεταρρυθμίσεων. Οι μεταρρυθμίσεις αυτές σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα πρέπει να είναι συντονισμένες προκειμένου να λάβουν υπόψη τους τις θετικές ή αρνητικές δευτερογενείς επιπτώσεις που μπορεί να έχουν από τη μία χώρα στην άλλη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε δύο νέες ανακοινώσεις το 2013 αναφέρεται στην ενδυνάμωση του χρηματοοικονομικού συντονισμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ιδιαίτερα στην Ευρωζώνη, σε ένα ψήφισμα το οποίο εγκρίθηκε σε 9 Δεκεμβρίου 2013, σε σχέση με τις ανακοινώσεις αυτές, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κάλεσε το Συμβούλιο να προχωρήσει σε πολιτικές δεσμεύσεις όσον αφορά την νομοθετική προετοιμασία που θα πρέπει να λάβει η χώρα για τις συνθήκες και την κοινοτική μέθοδο που θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για πιο καλά συντονισμένε οικονομικέ πολιτικέ στην Ευρωπαϊκή Ένωση και είπε ότι θα πρέπει να δοθούν επίση και να εγκριθούν κατευθυντήρε γραμμέ όσον αφορά την οικονομική σύγκληση των κρατών μελών και έχουν τεθεί από το Συμβούλιο συγκεκριμένοι περιορισμένοι στόχοι για τα πιο επίγοντα μέτρα. Επίσης, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καλεί εκ νέου τα κράτη-μέλη να διασφαλίσουν ότι τα εθνικά προγράμματα μεταρρύθμιση, τα οποία βαζίζονται στι κατευθύνε γραμμέ σύγκληση, θα πρέπει να συζητηθούν εκτενώς και να εγκριθούν και από τα εθνικά κοινοβούλια. Η συμμετοχή, η εμπλοκή των εθνικών κοινοβουλίων είναι πάρα πολύ σημαντική προκειμένου να καταφέρουμε να κάνουμε τα μέτρα αυτά πιο αποδεκτά από τους Ευρωπαίους πολίτες. Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο ψήφισμά μας αυτό λοιπόν του Δεκεμβρίου, λέμε ότι η κοινοβουλευτική αυτή διάσταση είναι πάρα πολύ σημαντική. Η διακοινοβουλευτική διάσκεψη που διοργανώθηκε από την Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων ήταν πάρα πολύ επικοδομητική. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοδομητική ανταλλαγή απόψεων που είχαμε και ελπίζουμε ότι ο πρόεδρος του ΕΚΟΦΗΝ θα καταφέρει πραγματικά να προωθήσει την δημοκρατική λογοδοσία στα πλαίσια της νέας οικονομικής διακυβέρνησης Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σας ευχαριστώ. Εγώ σας ευχαριστώ και δίνω το λόγο στην κυρία Περβάνς πρόεδρος της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κατά τη διάρκεια της διακοινοβουλευτικής συνάντησης που έγινε στα πλαίσια της Επιτροπής Απασχόλησης Κοινωνικών Υποθέσεων ασχοληθήκαμε με δύο θέματα. Το πρώτο αφορούσε την κοινωνική διάσταση της ΩΝΕ. Ε, πράγμα το οποίο μας επέτρεψε να θέσουμε τρία κύρια θέματα που μας απασχολούν. Το πρώτο αφορά το πόσο σημαντικές είναι οι κοινωνικές ανισορροπίες εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά κυρίως και εντός της ζώνης ευρώ. Πολλοί συνάδελφοι έλαβαν ε, τον ε, λόγο για να πούν ότι θα πρέπει εκτός από το θέμα των ανισοτήτων των μακροοικονομικών θα πρέπει να δούμε και τις κοινωνικές ανισορροπίες δεδομένου ότι θα μπορούσαμε να έχουμε επιπτώσεις ακόμη και σε αυτές τις ίδιες τις ανισορροπίες τις μακροοικονομικές. Κατά τη διάρκεια των συζητήσεών μας ένας Πολωνός συνάδελφος μας προειδοποίησε το ότι μία Ευρώπη πολλών ταχυτήτων και μία ε, πολιτική περιορισμένου περιθωρίου ελιγμών είναι κάτι το οποίο αποδυναμώνει την Ένωση και θα πρέπει κάθε κράτος να μπορέσει να κινητοποιηθεί ώστε τα θέματα τα κοινωνικά να τα λύσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Δεύτερο σημαντικό θέμα αφορούσε τον χάρτη πορείας και τους δείκτες έτσι όπως τους προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην ανακοίνωση του προηγουμένου Οκτωβρίου. Πολλοί παρεμβαίνοντος, κυρίως Ιρλανδοί, Γάλλοι, Ιταλοί και Έλληνες, έλαβαν το λόγο για να ζητήσουν, όπως έκανε στο ψήφισμα που ενέκρινε στην Ολομέλη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, οι δείκτες αυτοί να διευρυνθούν, ώστε να έχουμε ένα πλαίσιο περιορισμένο, πλην όμω να υπάρχουν περισσότεροι πλέον αυτών των πέντε που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για να μπορέσουμε να δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε το θέμα της ένδυας των παιδιών, των ε, καλών συνθήκων εργασίας και όλων των άλλων θεμάτων που αφορούν το δημογραφικό πρόβλημα. Τρίτο θέμα, το οποίο συζητήσαμε για την κοινωνική διάσταση της ε, πολιτικής, της οικονομικής και της ε, κοινωνικής είναι το θέμα του αυτόματου κοινωνικού απορριθμιστή. Αυτά είναι κάτι αποσταθεροποιητή. Πολλοί συνάδελφοι ανέφεραν αυτό το θέμα και είπαν ότι θα πρέπει με μία πρόταση που θα υποβάλουμε να μπορέσουμε να συμφιλιώσουμε τους πολίτες με την ε, συνεκτικότητα της κοινωνικής και οικονομικής ε, πολιτικής και της πολιτικής απασχόλησης ώστε να έχουμε ένα ελάχιστο ποσοστό επιδόματος ανεργίας ώστε να υπάρχει ένα ελάχιστο κατόφλι κοινωνικής προστασίας για τους πολίτες στα πλαίσια της ακρόασης που οργάνωσε την 9 ε, του Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο βάσει των πορισμάτων της μελέτης την οποία ζητήσαμε να γίνει και η οποία θα δημοσιευθεί στις 12 Φεβρουαρίου. Εκτός αυτών των τριών πυλώνων, αν θέλετε, των συζητήσεων που είχαμε, αναφέρθηκαν και διάφορα άλλα σημεία και βεβαίως η πρόκληση της ε, ανάπτυξης. Πολλοί συνάδελφοι ανέφεραν την διάσταση την κοινωνική και κυρίως πολλοί εξέφρασαν τις ανησυχίες, κυρίως ο Έλληνας συνάδελφος για την προοπτική μίας ανάπτυξης που θα θεωρηθεί ως ε, τριτοκοσμική και δεν θα είναι ανάλογη με αυτή στην οποία πρέπει να έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης, έγιναν ε, διάφορα σχόλια όσον αφορά τις προβλέψεις για πολύ μικρή ανάπτυξη που έκανε ο ΩΣΑ και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει προτείνει όπως ξέρουμε ανάλογα με κάθε τομέα μία ε, πολιτική ευφυή για να μπορέσουμε να έχουμε ανάκαμψη των επιπτώσεων δεδομένου ότι όπως βλέπουμε οι επενδύσεις ε, και η χρηματοδότηση σήμερα έχουν ε, μειωθεί. Επίσης, είπαμε ότι θα πρέπει να κάνουμε σε, σε θέματα κοινωνικής ευθύνης και περιβαλλοντική ευθύνη των εταιριών. Οι συνάδελφοι από τη Ρουμανία και τη Λετωνία υπενθύμησαν ότι η διαρθρωτική μεταρρύθμιση στην Ελλάδα επέτρεψε να καταπολεμήσουμε την ε, παράνομη εργασία, πράγμα το οποίο μας υπενθύμησε και ο υπεύθυνο Έλληνας Υπουργός, αλλά εκφράστηκαν ανησυχίες για τον ρυθμό που αναμένεται να δούμε όσον αφορά αυτές τις διορθωτικές μεταρρυθμίσεις. Εξετάστηκε ο ετήσιος ε, ρυθμός ανάπτυξης και ζητήθηκε να τονίσουμε κυρίως τον τρόπο με τον οποίο θα δοθούν εγγύησεις στους νέους. Και εδώ πρέπει να πω ότι υπάρχει κάτι το οποίο μας απογοήτευσε, διότι πολύ λίγες παρεμβάσεις έγιναν για αυτό το τόσο συγκεκριμένο θέμα, το οποίο μας κινητοποιεί βεβαίως όλους μόνο 17 κράτη-μέλη μέχρι σήμερα έχουν καταθέσει τα σχέδια ε, κινητοποίησης αυτής της εγκίνης προς τους νέους. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους Γάλλους και Ιταλούς συναδέλφους που μας εξήγησαν τι ακριβώς έγινε στις χώρες τους και με μεγάλη σαφήνεια είδα ότι πολλοί ενδιαφέρονται για την δημιουργία ενός δικτύου ώστε ο καθένας να συνεισφέρει με το τι ακριβώς κάνει στα πλαίσια αυτής της ευρωπαϊκής στρατηγικής και νομίζω ότι για όλους μας αυτό το θέμα ε, θα έχει μια προστιθέμενη ταξία για αύριο. Τώρα, γενικότερα, την αφορά τον ε, ρυθμό ετήσιας ανάπτυξης, τι διαπιστώνουμε. Πρώτα απ' όλα, ότι το 2014 και αναμφίβολα το 2015, λαμβάνοντας υπόψη τι προαναφέραμε για τις προβλέψεις που γίνονται και κυρίως εκ μέρους του Δουνουτού, ορισμένοι βλέπουν να επανέρχεται η ανάπτυξη, αλλά εύθραυστη ανάπτυξη και άνηση και μεταξύ κρατών μελών και μεταξύ των διαφόρων περιοχών εντός κάθε κράτους μέλους. Εκ παραλίλου, κάποια άλλη ανάπτυξη που μας απασχολεί είναι η ανάπτυξη και η ευάθυνση των, ανισοτήτων. Διότι στις ε, ε, αιτίες της κρίσης υπήρχαν και αυτές οι ανισότητες. Ανισότητες οι οποίες επιδεινώθηκαν από την ίδια την κρίση. Όσον αφορά τον ετήσιο έλεγχο των ε, ε, ανισοτήτων, πολλοί επανέλαβαν το γιατί οι εθνικές βουλές, το κοινοβούλιο και οι κοινωνικοί εταίροι δεν συμμετέχουν στην εξέταση αυτού του θέματος πρέπει να το κάνουν από κοινού και η Edith Bauer, συνάδελφος από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μας ανέφερε το θέμα των νέων χωρίς καμία εξειδίκευση. Και η συνάδελφος από την Σλοβακία μας είπε ότι αυτή τη στιγμή βλέπουμε ε, κάποιες πολιτικές οι οποίες γίνονται για την δημοσιονομική σταθερότητα να κατακερματίζουν και να καταστρέφουν το ανθρώπινο κεφάλαιο. Ήταν πάρα πολύ ε, πλούσιες οι συναντήσεις μας, δύο έγιναν και επέτρεψαν σε εκπροσώπους 12 εθνικών βουλών να παρέμβουν. Στην ε, τελευταία μας συνάντηση έλαβαν το λόγο 10 συνάδελφοι, μεταξύ των οποίων τέσσερις γυναίκες, συνάδελφοι. Είχαμε επίσης 12 παραμβαίνοντες στην πρώτη και τον Υπουργό και μεταξύ αυτών των 12 πάλι τέσσερις γυναίκες. Αυτά ήθελα να πω κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Και τώρα το λόγο έχει η κυρία Βέρτμαν, εκπρόσωπος του Προέδρου της Επιτροπής Προϋπολογισμού. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα Εν συντομία να σας παρουσιάσω τα συμπεράσματα της συζήτησής μας σχετικά με τη δημοσιονομική κατάσταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μιλήσαμε βεβαίως και για άλλα θέματα και για την πολιτική συνοχής και τονίσαμε πολλά χαρακτηριστικά της ε, πολιτικής αυτής και είπαμε ότι θα πρέπει να ενισχυθούν ε, πολλά στοιχεία της πολιτικής συνοχής η Ελλάδα, η Λιθουανία, η Ισπανία, η Σουηδία, η Πορτογαλία, εκπρόσωποι από τις χώρες αυτές πήραν το λόγο και μας μίλησαν για τις εμπειρίες τους ε, αλλά και για την σοβαρή κατάσταση στη χώρα τους. Από την Ελλάδα παραδείγματος χάρη ακούσαμε το τεράστια μείωση των θέσεων εργασίας και το τεράστιο ποσοστό της ε, ε, ανεργία των νέων που είναι κοντά στο 60%. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης των παρουσιάσεων το, από τους διάφορους ομιλητές κατέστησε φες ότι χρειάζονται μεγάλη υποστήριξη οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις για την προσπόρηση ε, κεφαλαίων, για την ανέβρεση κεφαλαίων. Πολλοί είπαν ότι υπήρξε στήριξη για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις αλλά τονίσαμε και τα, ε, το γεγονός ότι η πολιτική συνοχή είναι αυτή η οποία θα μπορούσε να στήριξει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και έτσι η είδαμε ότι με ένα πολύ μικρό κονδύλι που είχε δοθεί ουσιαστικά μέχρι τώρα πολύ μικρό ποσοστό 0,03% του ε, ΑΕΠ μπόρεσε να επιτευθεί ένα τα 100 ρυθμός ανάπτυξης μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι πολύ σημαντικό είναι πολύ σημαντική η στήριξη από εκεί και πέρα για τις επενδύσεις ακούσαμε τις χώρες που προανέφερα δεν ε, ε, γίνονται επενδύσεις, πράγμα που είναι ε, αρνητικό. Θα πρέπει λοιπόν να γίνουν κάποιες αλλαγές και όλοι είπαμε ότι πρέπει να επιδειχθεί μια κάποια ευελιξία για να μπορέσουν να προωθηθούν οι επενδύσεις. Εν ε, περιλήψη να πω ότι ότι ελέγχθη πως είναι πολύ περίπλοκοι οι κανόνες, υπάρχουν πάρα πολλές ιδιαιτερότητες στις διάφορες χώρες και ε, πράγμα το οποίο θα πρέπει να το προσέξουμε ιδιαίτερα. Οι επιστήμονες ουσιαστικά δεν έχουν χρόνο να ασχοληθούν με τα θέματα αυτά. Θα πρέπει όμως να γίνει προσπάθεια Παράδειγμα, ο, η μικρή ρυθμή απορρόφησης παραδείγματος χάρη ε, σε ορισμένες χώρες των ο, ε, κονδυλίων των ευρωπαϊκών. <coughs> Αυτό είναι ένα άλλο παράλληλο θέμα με τις επενδύσεις που θα πρέπει να μελετηθεί. Δημόσιες συμβάσεις. Αυτό ήταν ένα άλλο θέμα που ε, αναφέρθηκε και που, όπου δεν προχώρησαν τα πράγματα όσο έπρεπε και αυτό επηρεάζει βεβαίως και άλλες πτυχές. Ε, ελέγχθη επίσης ότι θα πρέπει να δοθεί μεγάλη σημασία στα, στην οροθέτηση για τα διάφορα προγράμματα και έργα. Το εκείνο το οποίο μας ενδιαφέρει είναι να είναι σαφής η στόχη των προγραμμάτων και των έργων που χρηματοδοτούνται εν μέρη λίγο ή περισσότερο από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, μιλήσαμε και λίγο για την απασχόληση δημιουργία θέσεων εργασίας αλλά τονίστηκε επίσης η ανάγκη για σωστή χρήση των κονδυλίων των διαρθρωτικών ταμείων των ευρωπαϊκών κονδυλίων και ε, η προσπάθεια που πρέπει να γίνει για μεγαλύτερη απορρόφησή τους. Ευχαριστώ πολύ. Εμείς ευχαριστούμε και τώρα το λόγο έχει ο Υπουργός Οικονομικών της Ελλάδος και πρόεδρος του ΕΚΟΦΗΝ, κύριος Γιάννης Τουρνάρας. Αξιότιμε Αντιπρόεδρε του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κύριε Κάρας, αξιότιμε Αντιπρόεδρε του Ελληνικού Κοινοβουλίου κύριε Τραγάκη, κυρίες και κύριοι μέλη του Ευρωπαϊκού και των Εθνικών Κοινοβουλίων. Με ιδιαίτερη χαρά και τιμή αποδέχθηκα την πρόσκληση του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κύριου Μάρτιν Σούλτς ε, προκειμένου να συμμετάσχω στην διακοινοβουλευτική διάσκεψη για την οικονομική διακυβέρνηση και το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο που οργανώθηκε από το Ευρωπαϊκό και το Ελληνικό Κοινοβούλιο. Ο θεσμός της Ευρωπαϊκής Κοινοβουλευτικής Ομάδας αποτελεί σημαντική ευκαιρία για ανταλλαγή απόψεων και αναζήτηση τρόπων ενίσχυσης της δημοκρατικής νομιμοποίησης στη διαδικασία λήψης των αποφάσεων και της συνεργασίας μεταξύ Ευρωπαϊκού και Εθνικών Κοινοβουλίων και αυτό αποδεικνύεται από τις συζητήσει που διεκθήσαν αυτό το τριήμερο. Για την ελληνική προεδρία, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μαζί με τα εθνικά κοινοβούλια θα είναι σημαντικοί εταίροι προκειμένου να ολοκληρωθούν οι στόχοι που έχουμε θέσει ως προτεραιότητες. Και αυτοί οι στόχοι είναι οι εξή. Πρώτον, προώθηση τη ανάπτυξη και απασχόληση στην Ευρώπη μέσω τη χρηματοδότηση τη πραγματική οικονομία. Η πρόσφατη οικονομική κρίση δημιούργησε σοβαρέ μακροοικονομικές ανισορροπίε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ευρωζώνη. Οι συνέπειε ήταν πολύ πιο έντονε στην περιφέρεια, με αποτέλεσμα να διευρυνθούν οι ανισορροπίε ανάμεσα στα κράτη-μέλη του πυρήνα και αυτών τη περιφέρεια. Παρ' όλα αυτά, η δημοσιονομική προσαρμογή και η εφαρμογή των διαθροτικών μεταρρυθμίσεων στα κράτη-μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση επέφεραν σημαντική διόρθωση στι εσωτερικέ και εξωτερικέ ανισορροπίε το έλλειμμα της γενικής κυβέρνησης περιορίστηκε, το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών μειώθηκε, ενώ οι προσαρμογές των μισθών και οι διαθροτικές μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας και προϊόντων οδήγησαν σε σημαντική βελτίωση της ανταγωνιστικότητας σε όρους κόστος εργασίας, ειδικά στα κράτη-μέλη που εντοπίζουν τα πιο σοβαρά προβλήματα. Παρ' όλα αυτά, απομένουν ακόμα πολλά να γίνουν. Η ανεργία και η φτώχεια παραμένουν σε υπερβολικά υψηλά επίπεδα και η πολιτική μας θα πρέπει να επικεντρωθεί στην αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών που επηρεάζουν μεγάλο αριθμό Ευρωπαίων πολιτών. Τόσο το ιδιωτικό όσο και το δημόσιο χρέο έχουν σταθεροποιηθεί σε σχετικά υψηλά επίπεδα παρά τι προσπάθειε που καταβάλλονται. Οι πλεονασματικέ χώρε θα χρειαστεί να προσπαθήσουν ακόμα περισσότερο για τη στήριξη τη εγχώρια ζήτηση. Οι μακροοικονομικέ ανισορροπίε διαφέρουν από χώρα σε χώρα. Θα πρέπει όμω να δώσουμε προσοχή σε όλε τι περιπτώσει ανεξάρτητα από το εάν πρόκειται για πλεονασματικέ ή ελληνικέ χώρε. Η ελληματικε χωρες Επιτροπή δημοσίευσε τον Νοέμβριο του 2013 την έκθεση μηχανισμού επαγρύπνηση, δηλαδή το Alert Mechanism Report, η οποία έκθεση επισημαίνει τα κύρια πεδία ανισορροπιών για κάθε χώρα. Πιστεύουμε ότι η άσκηση αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική και ενθαρρύνουμε όλα τα κράτη-μέλη να λάβουν σοβαρά υπόψη τις συστάσεις της έκθεσης αυτής η ελληνική προεδρία αναγνωρίζει τη σημασία της έκθεσης και θα βασιστεί σε αυτήν για την προετοιμασία των συμπερασμάτων του Συμβουλίου Οικονομικών και Δημοσιονομικών Υποθέσεων, δηλαδή του ΕΚΟΦΗΝ, του Φεβρουαρίου. Ένα άλλο σημαντικό εργαλείο είναι οι εμπεριστατωμένες επισκοπήσεις, δηλαδή τα in-depth reviews, οι οποίες θα εξετάσουν σε μεγαλύτερο βάθος τις μακροοικονομικές ανισορροπίες που επισημάνθηκαν στην έκθεση μηχανισμού επαγρύπνησης για κάθε κράτος μέλος και θα προτείνουν τις κατάλληλες συστάσεις πολιτικής η ελληνική προεδρία στηρίζει την όλη διαδικασία και παίρνει τις απαραίτητες πρωτοβουλίες για την επιτυχή διεξαγωγή της άσκησης αυτής. Τέλος, θα ήθελα να σας ενημερώσω για την πρόοδο που έχει σημειωθεί τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα όσον αφορά τη διόρθωση των ανισορροπιών. Η Ελλάδα, όπως ξέρετε, υπέφερε από μεγάλες και διαρκείς ανισορροπίες. Το 2008 το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεξών συναλλαγών ήταν 14,9% του ΑΕΠ. Το 2014 προβλέπεται πλεόνασμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών της τάξης του 1,3% του ΑΕΠ. Μεταξύ του 2009 και του 2013 το έλλειμμα της γενικής κυβέρνησης μειώθηκε κατά 13,4 εκατοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ, δηλαδή από μείον 15,6% σε μείον 2,2%. Επίσης, το πρωτογενές έλλειμμα μειώθηκε κατά 10,8 εκατοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ, από έλλειμμα της τάξης του 10,4% σε πλεόνασμα της τάξης του 0,4%. Και συγγνώμη που σας απασχολώ με τόσα νούμερα, αλλά θέλω να τονίσω ότι πρόκειται για τη μεγαλύτερη και γρηγορότερη προσαρμογή που έχει καταγραφεί ποτέ σε οικονομία του ΩΣΑ. Ενώ το κυκλικά διορθωμένο πρωτογενέ πλεόνασμα, που σύμφωνα με όλου του οικονομολόγου πρέπει να είναι ο δείκτη στον οποίο πρέπει να προσέχουμε, αναμένεται να ξεπεράσει το 6% του ΑΕΠ σχετικά με το θέμα της χρηματοδότησης της οικονομίας για την τόνωση της ανάπτυξης και της απασχόλησης που αποτέλεσε αντικείμενο ενδιαφέροντος της χθεσινής ημέρας θα ήθελα να τονίσω ότι για την ελληνική προεδρία αποτελεί κεντρική προτεραιότητα. Η Ευρώπη εξακολουθεί να κινείται σε τροχιά δημοσιονομικής εξυγίανσης και τα πρώτα σημάδια ανάκαμψης είναι ήδη ορατά. Τα ποσοστό ανεργίας έχουν σταθεροποιηθεί, αν και ανήλθανε σε ανεπίτρεπτα υψηλά επίπεδα στις χώρες εκείνες που εφαρμόζουν προγράμματα προσαρμογής η ευρύτερη κοινωνική κατάσταση εξακολουθεί να είναι δύσκολη. Για τον λόγο αυτό προβάλλει επιτακτική ανάγκη να επικεντρώσουμε τις πολιτικές μας στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και παράλληλα στην τόνωση της επιχειρηματικότητας. Διότι μόνη της, από μόνη της μάλλον, η δημοσιονομική προσαρμογή χωρίς παράλληλες πολιτικές φιλικές προς την ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή μετατρέπεται σε παραταταμένη λιτότητα η οποία αποξενώνει τους πολίτες και τους οδηγεί και οδηγεί σε ενίσχυση του ευρωσκεπτικισμού. Βασική προϋπόθεση για την επιστροφή στην ανάπτυξη και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας είναι η ομαλή ροή χρηματοδότησης της οικονομίας. Η οικονομική κρίση προκάλεσε πρωτοφανή πτώση στις επενδύσεις σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου εξακολουθούν να είναι περίπου 17% χαμηλότερες από το ανώτατο όριο που επετεύχθη το 2008 Μάλιστα, στι χώρε που επλήγησαν περισσότερο από την κρίση, όπω είναι η Ελλάδα, η Ιρλανδία, η Πορτογαλία, η Ισπανία και η Κύπρο, το ποσοστό μείωση είναι ακόμα μεγαλύτερο, περίπου 40 με 50% κάτω. Η χρηματοδότηση τη ευρωπαϊκή οικονομία βασίστηκε σε πολύ μεγάλο βαθμό στην τραπεζική διαμεσολάβηση. Αυτό επέφερε σημαντική μείωση στη διαθεσιμότητα τραπεζική μακροπρόθεσμη πίστη κατά την περίοδο τη κρίση που ακολούθησε. Αποτέλεσμα των παραπάνω, ήταν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της ευρωπαϊκής οικονομίας όχι μόνο του ευρωπαϊκού νότου αλλά όλης της ευρωπαϊκής οικονομίας να πληγούν περισσότερο. Η έλλειψη ρευστότητας ομολογουμένως συντέλεσε στη διαιώνιση της κρίσης. Δυστυχώς αυτή η παράμετρος δεν ελήφθη σοβαρά υπόψη όσο θα έπρεπε για την εξήγηση πολλών φαινομένων κατά τη διάρκεια αυτής της δύσκολης περίοδου. Η οικονομική και πολιτική αβεβαιότητα υπήρξαν βασικοί αποτρεπτικοί παράγοντες στην προσέλκυση νέων επενδύσεων στην Ευρωζώνη κατά τη διάρκεια της κρίσης. Όσο δυσάρεστο και αν είναι αυτό, οφείλω να αναφερθώ σε ατυχείς δηλώσεις πολλών παραγόντων, ακόμα και μέσα στην Ευρωζώνη, που δεν απέφυγαν αναφορές στον ενδεχόμενο εξόδου από το ευρώ. Παράλληλα με την ενίσχυση των κλασικών τραπεζικών πηγών χρηματοδότηση, θα πρέπει να αναζητήσουμε και εναλλακτικέ πηγέ πρόσβαση των επιχειρήσεων σε ρευστότητα. Κατ' εφαρμογή των συμπερασμάτων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, η Προεδρία θα συνδράμει το Συμβούλιο ΕΚΟΦΗΝ στην παρακολούθηση τη πορεία εξέλιξη των εργαλείων για τη χρηματοδότηση τη οικονομία και ιδιαίτερα τη διευκόλυνση τη πρόσβαση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση με στόχο την ενίσχυση τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασία η ελληνική προεδρία θα προωθεί στο διάλογο βάσει μια σειρά δράσεων που αναμένεται να προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε συνέχεια τη Πράσινη Βίβλου σχετικά με τη μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση τη οικονομία και τη διευκόλυνση τη πρόσβαση των μικρομεσαίων των επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση. Στο πλαίσιο αυτό, η Προεδρία μα θα επιταχύνει τι συζητήσει για τη χρηματοδότηση τη ανάπτυξη με βάση τι συστάσει τη ομάδα εμπειρογνωμόνων υψηλού επίπεδου κατ' εφαρμογή της εξιοδότησης του άτυπου Συμβουλίου ΕΚΟΦΗΝ στι 12 Απριλίου 2013. Η Ελληνική Προεδρία χαιρετίζει τη νέα εντολή τη Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων για αύξηση της χρηματοδότησης των δραστηριοτήτων του και θα υποστηρίξει την Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα των Επενδύσεων στι προσπάθειέ του για περαιτέρω ενίσχυση των δυνατοτήτων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων, με την αύξηση των κεφαλαίων του και με σκοπό την επίτευξη τελική συμφωνία μέχρι το Μάιο του 2014 η συγκεκριμένη απόφαση θα αποτελέσει ένα ακόμα βήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την αποκατάσταση της κανονικής δανειακής ροής προς την οικονομία. Η διαδικασία προβλέπει συναπόφαση του Κοινοβουλίου και ευελπιστούμε να υπάρξει γρήγορα συμφωνία επί της πρότασης. Τέλος, σε επίπεδο νομοθετικών πρωτοβουλειών, σημαντικός θεωρείται ο κανονισμός για τα μακροπρόθεσμα επενδυτικά κεφάλαια, ο οποίος συνδέεται με τη χρηματοδότηση έργων υποδομών και την ανάπτυξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Θα μου επιτρέψετε να πάω τώρα στο δεύτερο μεγάλο στόχο, που είναι η ενισχυμένη δημοσιονομική εποπτεία και η ενισχυμένη γονικότερα αρχιτεκτονική της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης. Η πρόσφατη οικονομική κρίση κατέδειξε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ευρωζώνη έπρεπε να ενισχύσουν το συντονισμό και τη συνεργασία τους στο σχεδιασμό της δημοσιονομικής τους πολιτικής και να λάβουν όλα τα απαραίτητα διορθωτικά μέτρα στην περίπτωση που αυτό χρειαστεί. Η ανάγκη για περαιτέρω συντονισμό οδήγησε στην εισαγωγή του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, του ημερολογίου δηλαδή, για την χάραξη πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Ευρωπαϊκό Εξάμενο μέχρι στιγμής υπήρξε επιτυχές ιδιαίτερα αν ληφθεί υπόψη ότι η οικονομική κατάσταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ιδιαίτερα στα κράτη-μέλη που έχουν πληγεί περισσότερο από την οικονομική κρίση έχει βελτιωθεί σημαντικά. Οι ενισχυμένοι κανόνε για την οικονομική διακυβέρνηση, δηλαδή το εξάπτυχο, το six-pack, το δίπτυχο, το two-pack και η συνθήκη για τη σταθερότητα, το συντονισμό και τη διακυβέρνηση εφαρμόζονται πλήρω σε αυτόν τον κύκλο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και η επιτυχή ολοκλήρωσή του αποτελεί κύρια προτεραιότητα τη Ελληνική Προεδρία. Μετά την παρουσίαση τη έκθεση προ μια ουσιαστική οικονομική και νομισματική ένωση στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Δεκεμβρίου του 2012, προχώρησαν οι εργασίε επάνω στα βασικά συστατικά στοιχεία για την ενδυνάμωση τη αρχιτεκτονική οικονομική και Νομισματικής ένωση. Στο πλαίσιο αυτό, η ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ένωσης είναι ουσιώδης για την αποκατάσταση της αξιοπιστίας του χρηματοπιστωτικού μας τομέα και την εξασφάλιση της λειτουργίας του προ όφελο της πραγματικής οικονομίας, προ όφελο των επιχειρήσεων που επιθυμούν να προβούν σε παραγωγικέ επενδύσει και να δημιουργήσουν θέσει απασχόληση, προ όφελο τέλο των ε, σκληρά εργαζόμενων νοικοκυριών που αποταμιεύουν για ένα καλύτερο μέλλον. Η Τραπεζική Ένωση είναι απαραίτητη ώστε να σπάσει οριστικά ο φαύλο κύκλο μεταξύ των τραπεζών και του δημόσιου χρέου που βρίσκεται στο επίκεντρο τη χρηματοπιστωτική κρίση. Χρειαζόμαστε επίση την Τραπεζική Ένωση ώστε να εξασφαλιστούν οι κατάλληλες εκείνες συνθήκες για τη διατήρηση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας στην οποία βασίζονται η ευημερία των επιχειρήσεων και η προστασία των καταθέσεων. Εκτός από την προώθηση της Τραπεζικής Ένωσης, οι συζητήσεις για την εμβάνθηση της ΟΝΕ, της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης, έχουν επικεντρωθεί στον εκ των προτέρων συντονισμό των κύριων οικονομικών μεταρρυθμίσεων, στην κατάρτιση εταιρικών σχέσεων για την ανάπτυξη, την απασχόληση και την ανταγωνιστικότητα, καθώς και στην κοινωνική διάσταση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης. Για πρώτη φορά, η κοινωνική διάσταση της ΟΝΕ θα ενσωματωθεί στον κύκλο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου για το 2014. Η Ελληνική Προεδρία, υλοποιώντα τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, θα επιδιώξει να διευκολύνει περαιτέρω τι συζητήσει για την εξέλιξη τη Οικονομικής και Ένωση. Τέλο, ο τρίτο στόχο. Ποιε είναι οι προτεραιότητε για τον κύκλο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου για το 2014. Το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο δημιουργεί ένα σημαντικό πλαίσιο για στενότερη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών για το συντονισμό της οικονομικής πολιτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ελληνική Προεδρία θα βασιστεί στην εμπειρία των προηγούμενων ετών, ιδιαίτερα στην πολύ καλή διαχείριση της Ιρλανδικής Προεδρίας, για να ολοκληρώσει αυτή τη διαδικασία με τη μέγιστη δυνατή επιτυχία η ελληνική προεδρία θα εστιάσει στην αποτελεσματική εφαρμογή των δεσμεύσεων που απορρέουν τόσο από το δημοσιονομικό σύμφωνο όσο και από το ενισχυμένο σύμφωνο σταθερότητα και ανάπτυξη. Φέτο, το Ευρωπαϊκό Εξάμενο παρουσιάζει τέσσερι καινοτομίε. Διευρυμένο ρόλο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στην καθοδήγηση τη όλη διαδικασία. Διαφοροποίηση στη συμμετοχή των συνθέσεων του Συμβουλίου σε συνέχεια των συστάσεων από τα διδάγματα της μέχρι σήμερα διαδικασίας, οι συζητήσεις του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου θα πραγματοποιούνται μόνο στα τομεακά συμβούλια, όπου μια τέτοια συζήτηση φέρνει σαφή προσθέμενη αξία. Εφαρμογή των ειδικών αναχώρα συστάσεων, δηλαδή των Country Specific Recommendations. Το νέο παράρτημα της ετήσιας επισκόπησης της ανάπτυξης, δηλαδή το Annual Growth Survey, επικεντρώνεται στην υλοποίηση των ειδικών συστάσεων αναχώρα από τα κράτη-μέλη το Συμβούλιο αναμένεται να δώσει μεγαλύτερη προσοχή στον τρόπο που τα κράτη-μέλη θα εφαρμόσουν αυτές τις συστάσεις. Το χρονοδιάγραμμα για την έγκριση των ειδικών αναχώρας συστάσεων, των CSRs, αποτελεί μια επιπλέον πρόκληση για την Προεδρία μας, καθώς θα κληθούμε να διαχειριστούμε αυτή τη διαδικασία μέσα σε σχετικά στενά χρονικά περιθώρια. Για τον λόγο αυτό εργαζόμαστε προκειμένου να ολοκληρωθεί η όλη διαδικασία όσο το δυνατό πιο έγκαιρα και αποτελεσματικά. Είμαστε σε στενή επαφή με την Επιτροπή και τους Προέδρους των Αρμόδιων Επιτροπών που επεξεργάζονται τις ειδικέ αναχώρα ε, συστάσεις μετά τη δημοσίευσή τους από την Επιτροπή προκειμένου να εξασφαλίσουμε την αποτελεσματική εποπτεία της όλης διαδικασίας. Όλα τα κράτη-μέλη είναι σύμφωνα με τις πέντε γενικές προτεραιότητες που επισημάνθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης, δηλαδή την επιδίωξη δημοσιονομικής εξυγίανσης φιλικής ε, προς την ανάπτυξη, την αποκατάσταση της ροή των δανείων στην οικονομία, την προώθηση της ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας για το σήμερα και το αύριο, την αντιμετώπιση τη ανεργία και τέλο, τον εξυγχρονισμό τη δημόσια διοίκησης. Η Ελληνική Προεδρία θα επικεντρωθεί σε αυτέ τι προτεραιότητε κατά τη διάρκεια τη όλη διαδικασία του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Ειδικότερα, το ΕΚΟΦΗΝ, δηλαδή το Συμβούλιο Οικονομικών και Δημοσιονομικών Υποθέσεων του Φεβρουαρίου, θα υιοθετήσει συμπεράσματα τα οποία θα υποβληθούν στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Μαρτίου και τα οποία θα παρέχουν καθοδήγηση για την εφαρμογή των προτεραιοτήτων που συμφωνήθηκαν στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Δεκεμβρίου του 2013 για μακροοικονομικά και δημοσιονομικά θέματα, καθώ και συμπεράσματα για την έκθεση του Μηχανισμού Επαγρύπνηση. Μετά την υιοθέτηση των εμπεριστατωμένων επισκοπήσεων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Συμβούλιο ΕΚΟΦΗΝ του Μαΐου θα υιοθετήσει τα σχετικά συμπεράσματα. Τέλος, το Συμβούλιο ΕΚΟΦΗΝ του Ιουνίου θα υιοθετήσει τη γνώμη του Συμβουλίου για τις ειδικέ αναχώρασης στάσεις, ώστε να εγκριθούν από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ε, του Ιουνίου. Σας ευχαριστώ πολύ. Εμείς ευχαριστούμε τον Έλληνα Υπουργό των Οικονομικών και το λόγο έχει ο κύριος Δημήτριος Κερμαστινός, βουλευτής από την Ελλάδα. Έχετε το λόγο. Ε, κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να σχολιάσει περισσότερο ε, ο κύριος Τουρνάρας ε, το θέμα που συζητήσαμε χθες με επευκαιρία της ερώτησης των όλοι Ρεν. Ότι δηλαδή <clears throat> με το να ε, διαβεβαιώνει ότι οι τράπεζες, η Κεντρική Τράπεζα εγγυάται τα 100.000 ευρώ σαν όριο για τους καταθέτες υπό την έννοια ότι δηλαδή δεν θα γίνει ένα haircut των καταθετών στις τράπεζες αυτό στην ουσία ενισχύει τις ε, κεντρικές τράπεζες, τις τράπεζες των βορείων χωρών που είναι ισχυρότερες γιατί ήδη από τον Νότο και ιδιαίτερα από την Ελλάδα υπάρχουν καταθέσεις προς τις τράπεζες αυτές της τάξεως των 50 με 60 δισεκατομμυρίων όπως υπολογίζεται. Και το ερώτημα είναι πώς μπορεί οι τράπεζες αυτές να εγγυηθούν την ανάπτυξη, δηλαδή να χορηγήσουν δάνεια σε επιχειρήσεις μικρομεσαίες, ούτως ώστε να γίνει ανάπτυξη. Διότι εάν δεν συμβεί με αυτόν τον τρόπο η ανάπτυξη, ο δεύτερος τρόπος είναι ε, με τους επενδυτές οι οποίοι βέβαια επενδυτές πολύ φυσικό περιμένουν να υπάρχει μια αγορά πολύ έτσι επικερδής για αυτούς όπως είναι οι αγορές των τρίτων χωρών που αν αυτό συμβεί για τις χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου τότε θα έχουμε πια πραγματικά δύο ταχύτητες ανάπτυξης της ανάπτυξης των χωρών της Ευρώπης του Βορρά και του τριτοκοσμικού Νότου όπως θα εξελιχθεί τριτοκοσμικός Νότος και βεβαίως ε, η ερώτηση αυτή είχε απευθυνθεί στον Όλι Ρεν ο οποίος ε, από ό,τι είδατε χθε δεν την σχολίασε, δεν την απήντησε. Τώρα σήμερα η ερώτηση δεν είναι προς εσάς αλλά είναι εμέσως προς εσάς ότι υπό την έννοια ότι πρέπει ε, τελικά να εξασκηθεί κάποια πίεση ε, προς αυτή την κατεύθυνση ούτως ώστε να υπάρχει τουλάχιστον ίση συμπεριφορά όσον αφορά τους καταθέτες και στις τράπεζες του Βορρά και στις τράπεζες του Νότου. Ε, ε, αντιλαμβάνομαι ότι είναι δύσκολο εσείς να το σχολιάσετε αλλά ε, αντιλαμβάνεστε ότι είναι ένα ζωτικό θέμα για την ανάπτυξη των χωρών του Νότου και ειδικότερα της Ελλάδας όταν αυτό το, το θέμα κατά κάποιο τρόπο επισκιάζεται σαν συνεφιά. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Κρεμαστινό. Και τώρα το λόγο έχει ο κύριος Μαρινή, πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων της Γαλλικής Γερουσίας. Oui, Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, τη στιγμή για την οποία ολοκληρώνεται αυτή η συνάντηση, θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι θα πρέπει να σημειώσουμε πρόοδο όσον αφορά τον τρόπο λειτουργίας και το καθεστώς που διέπει αυτή τη διακοινοβουλευτική συνέλευση. Συγγνώμη που επαναλαμβάνομαι, αλλά τα συμπεράσματα του Βίλνους δεν υλοποιήθηκαν πλήρως δεδομένου ότι προβλεπόταν να δημιουργηθεί μια ομάδα εργασίας για να ορίσει τον τρόπο λειτουργίας αυτής της διάσκεψης. Η ομάδα αυτή εργασίας έως σήμερα δεν συνεδρίασε και από όσον κατάλαβα θετικό είναι αυτό. Στο χρονοδιάγραμμα των επομένων μηνών προβλέπει η Ελληνική Προεδρία, αλλά κυρίως η προπαρασκευή της Ιταλικής Προεδρίας θα θέσουν επιτάπητος το θέμα αυτό και πάλι. Επιτρέψτε μου να πω ότι μία διακοινοβουλευτική διάσκεψη η οποία θα ελέγχεται υπερβολικά από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν είναι μια διακοινοβουλευτική διάσκεψη έτσι όπως προβλέπεται στο άρθρο 13 της συνθήκης που είναι η βάση μας και θα πρέπει να είναι δυνατόν χωρίς να διαταράξουμε την ισορροπία των θεσμικών μας οργάνων να αποδεχθούμε το ότι μπορούμε σε συνεννόηση με εκπροσώπους των ενδιαφερομένων ε, επιτροπών των Εθνικών Βουλών να ετοιμάσουμε αυτές τις συνεδριάσεις, τις εξαμηνίες, να καθορίσουμε ένα τρόπο λειτουργίας με τη συνδρομή της γραμματείας και να εξασφαλίσουμε το ότι όλα αυτά θα είναι μια συνεχιζόμενη διαδικασία. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο βεβαίως του οποίου η θητεία λύγει σε λίγους μήνες, καλό θα ήταν να μας βοηθήσει να το κάνουμε κάτι τέτοιο σε ένα πνεύμα, εάν ε, θέλετε, πιο καλή συνεργασία στα πλαίσια του τέλους της παρούσας θητείας. Ξέρουμε ότι βεβαίως Προβλέπονται οι ευρωεκλογέ, υπάρχει μεγάλη κινητικότητα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και μπορούμε να θεωρήσουμε ότι θα εφαρμοστεί πλήρως το άρθρο 13. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον κύριο Μαρινή και το λόγο το έχει τώρα η κυρία Τίσεν, Ευρωβουλευτή. Eh, eh, eh, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ο πρόεδρος του, ο προεδρεύων μάλλον του ΕΚΟΦΗΝ πολύ σωστά μας είπε ότι θα πρέπει να προωθηθεί ιδιαίτερα η Τραπεζική Ένωση του ώστε να επανέλθει η εμπιστοσύνη των πολιτών. Ξέρουμε πολύ καλά ότι ε, η εμπιστοσύνη αυτή έχει εκλείψει, έχει μειωθεί τώρα τελευταία. Έχουμε ε, κάποιους κανονισμούς βεβαίως, έχουμε κάποιους κανόνες, έχουμε το σύστημα εποπτείας, υπάρχουν όλα αυτά ήδη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά ο, ο μηχανισμός η MSR είναι ακόμη κατά την άποψη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πολύ πιο περίπλοκος και γι' αυτό δεν βοηθάει τα πράγματα. Γι' αυτό ε, που φαντάζεται κανείς μια διακρατική λύση και ενδεχομένως ίσως όχι μια κοινή λύση. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω τον ε, Έλληνα Υπουργό αν πιστεύει ότι θα μπορέσουμε τελικά να φτιάξουμε έναν ενιαίο ομοιόμορφο ενιαίο ευρωπαϊκό μηχανισμό για όλους γιατί μας χρειάζεται αυτό για την Τραπεζική Ένωση αυτό είναι το βασικό σημείο Το λόγο έχει ο κύριος από το Βελγικό Κοινοβούλιο σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ ιδιαίτερα για τη διοργάνωση αυτής της κοινοβουλευτικής διάσκεψης. Είναι πάρα πολύ σημαντικό εκπρόσωποι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των Εθνικών Κοινοβουλίων να συναντιόνται και να μιλάνε, μόνο ότι μπορεί να μην συμφωνούμε πάντα για τον τρόπο εργασίας, για τη μέθοδο εργασίας. Το είπε αυτό και ο κύριος Μαρινή και δεν προσεγγίσουμε πάντα τα πράγματα από την ίδια οπτική γωνία, από την ίδια σκοπιά. Ωστόσο πρέπει να σας πω ότι η διάσκεψη αυτή από μόνη τη δεν επαρκεί όσον αφορά την δημοκρατική πρόκληση που έχουμε μπροστά μας, το ότι θα πρέπει δηλαδή οι Ευρωπαίοι πολίτες να συνειδητοποιήσουν όλο και περισσότερο ότι είναι χρήσιμο το ευρωπαϊκό οικοδόμημα, ότι είμαστε πεπισμένοι γι' αυτό. Βλέπουμε ότι υπάρχουν συγκεκριμένοι κανόνε στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου που μπορούν να επηρεάσουν πάρα πολύ σημαντικά τα κράτη-μέλη. Υπάρχουν λοιπόν κάποια πράγματα τα οποία ακόμα πρέπει να βελτιωθούν και να διορθωθούν. Θα πρέπει να καταφέρουμε να εμπλέξουμε περισσότερο του ε, κοινωνικού εταίρους στου μηχανισμού σύγκληση που έχουμε επιτάπητος σήμερα και θα πρέπει επίσης να είμαστε πολύ προσεκτικοί όσον αφορά τις ιδιαίτερότητε των επιμέρους κρατών μελών. Τώρα από οικονομικής πλευράς τα οικονομικά μέτρα τα οποία έχουν επιβληθεί στα κράτη-μέλη, εκ των οποίων ορισμένα θα επιστρέψουν σε οικονομική ανάκαμψη, ουσιαστικά έχουν οδηγήσει κυρίως σε ύφεση, με έντονες κοινωνικές επιπτώσεις, τις οποίες υπενθύμησε η κυρία Μπερές, καθώς επίσης και οι υπόλοιποι συμμετέχονται στην ομάδα εργασίας της σήμερα το πρωί. Αύξηση δηλαδή της ένδυας, αύξηση επίσης της ανισότητος μεταξύ των πολιτών των κρατών μελών, Καταλαβαίνετε ότι δεν μπορούμε να εργαστούμε κατά τρόπο κατακαιρματισμένο όσον αφορά τα κοινωνικά αυτά ζητήματα. Έχουμε την τύχη να έχουμε σήμερα μαζί μας ε, τον ε, Προεδρεύοντα του ΕΚΟΦΗΝ. Θα ήθελα λοιπόν να πω προς τον Προεδρεύοντα του ΕΚΟΦΗΝ ότι ε, ενδιαφερόμαστε ιδιαίτερα για όλα αυτά τα νέα μέτρα τα οποία θα πρέπει να εγκρίνουμε. Και πέρα από το μηχανισμό εξυγίανση, θα πρέπει να καταφέρουμε να αποφύγουμε μια επόμενη μελλοντική τραπεζική κρίση. Θα πρέπει ο τραπεζικός τομέας να δραματίσει το ρόλο του, δηλαδή τη χρηματοδότηση της οικονομίας. Θα πρέπει να ασχοληθούμε με το ζήτημα αυτό, καθώς επίσης και μετά όσα προβλέπει η έκθεση Λίκανεν όσον αφορά τη διαφοροποίηση των διαφορετικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Θα έχουμε τη δυνατότητα να ανταλλάξουμε απόψεις και στις επόμενες συναντήσεις που θα έχουμε εξ ονόματο Ευρωπαϊκή Επιτροπή και του Συμβουλίου, εκ μέρου μάλλον τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και του Συμβουλίου, θα θέλαμε ένα οικονομικό κοινωνικό συμβούλιο το οποίο να λαμβάνει υπόψη του επίση και τα ενεργειακά θέματα τα οποία πολλές φορές βρίσκονται στο περιθώριο. Νομίζω ότι ε, όσον αφορά την κλιματική αλλαγή και όσον αφορά τα οικονομικά ζητήματα υπάρχουν ε, πάρα πολλές θέσεις απασχόλησης που θα μπορούσαν να δημιουργηθούν στα πλαίσια των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της ενεργειακής αποδοτικότητος. Θεωρώ λοιπόν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να εκμεταλλευτεί τη χρυσή αυτή ευκαιρία και να ασκήσει πίεση στα κράτη-μέλη προκειμένου να ακολουθήσουν αυτό το δρόμο. Σας ευχαριστώ πολύ. Εμείς ευχαριστούμε και τώρα το λόγο έχει ο κύριος Δημήτρης Παπαδημούλης βουλευτής από την Ελλάδα και αντιπρόεδρος της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Στουρνάρα, χθε ο επικεφαλής του Eurogroup, ο κύριος Ντάισεμπλουμ, είπε ότι δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί πότε θα επιστρέψει η Τρόικα στην Αθήνα, γιατί με ευθύνη της ελληνικής κυβέρνησης δεν έχουν υλοποιηθεί κάποια προαπαιτούμενα. Δέκα μέρες νωρίτερα ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο κύριος Σαμαράς, μιλώντας στο Ευρωκοινοβούλιο στο Στρασβούργο, είπε το περίφημο «We delivered». Η ελληνική κυβέρνηση τα έχει κάνει όλα. Ποιος λέει την αλήθεια από τους δυο. Εσείς είπατε ότι δεν σας πολύ απασχολεί και πότε ακριβώς θα γυρίσει η Τρόικα. Μπορείτε να μας πείτε στο συγκεκριμένο θέμα τι πιστεύει η ελληνική κυβέρνηση. Υπάρχουν εκκρεμότητες και ποιες. Θέλετε να γυρίσει η Τρόικα στην Αθήνα και πότε. Δεύτερη ερώτηση και παρακαλώ απαντήσεις όσο δυνατόν πιο συγκεκριμένες. Η έκθεση, το σχέδιο έκθεσης Επιτροπής του Ευρωκοινοβουλίου θεωρεί ότι υπάρχει ένα μεγάλο έλλειμμα δημοκρατικής νομιμοποίησης και διαφάνειας στο πώς δούλεψε και δουλεύει η Τρόικα και στην Ελλάδα και στις άλλες χώρες. Ποια είναι η δική σας γνώμη ως ελληνική προεδρία. Υπάρχει θέμα δημοκρατίας και διαφάνειας ή όχι. Τρίτο θέμα η γνωμοδότηση Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων του Ευρωκοινοβουλίου εκτός από τη δημοσιονομική προσαρμογή για την οποία μας μιλήσατε σημειώνει και το ρεκόρ ύφεσης και το ρεκόρ ανεργίας και το ρεκόρ φτώχειας και μιλά για τις τεράστιες κοινωνικές επιπτώσεις τις καταστροφικές από την εφαρμογή του μνημονίου και στην Ελλάδα και στις άλλες χώρες. Ποια είναι η γνώμη της ελληνικής προεδρίας γι' αυτά. Και τέλος, είναι φανερό πια από τους αριθμούς ότι το χρέος που αυξήθηκε στα χρόνια του μνημονίου και στην Ελλάδα και στις άλλες χώρες και σε όλη την Ευρωζώνη είναι ένα ευρωπαϊκό πρόβλημα και όχι μόνο ένα πρόβλημα του Νότου που επιτείνει τις ανισορροπίες και απειλεί και τις οικονομίες και τις κοινωνίες και το ίδιο το νόμισμα. Πώς θα αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα κατά τη γνώμη σας και πότε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Αντιπρόεδρε, κύριε Υπουργέ, άκουσα με μεγάλη προσοχή τις προτεραιότητες της ελληνικής προεδρίας στι ε, στις οποίες αναφερθήκατε και θέλω να πω καταρχάς πόσο φυσικά ένα ε, ε, ισορροπημένο και ολοκληρωμένο σχέδιο αλλά θέλω να πω πόσο σημαντικό θεωρώ ότι λέτε καθαρά και συγκεκριμένα και στοχευμένα την ανάγκη ε, χρηματοδότησης της πραγματικής οικονομίας και την υποστήριξη των εναλλακτικών μέσων. Θα έχουμε τη δυνατότητα, ενώ εναλλακτικών πέρα από το τραπεζικό σύστημα, το οποίο υποφέρει παντού, ε, θα έχουμε την ευκαιρία και το απόγευμα στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων να το συζητήσουμε. Ε, αναφερόμενοι στο χρέος, στο δημόσιο χρέος, κύριε Υπουργέ, είναι ένα θέμα για την χώρα μας και ένα στόχος πολιτικός η βιώσιμη αντιμετώπιση του. Αλλά κύριε Υπουργέ, ε, ως Προεδρεύον του ΕΚΟΦΗΝ έχετε κατά νου κάποια πρωτοβουλία γιατί είναι ένα ευρωπαϊκό ε, παγκόσμιο πρόβλημα το θέμα του χρέους που απειλεί την ανάπτυξη και τη σταθερότητα. Έχει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ξέρω ότι παρακολουθείτε τις εκθέσεις μας, τις απόψεις μας, έχει πολλές φορές εκφραστεί, έχει εκφράσει, ε, προτείνει ε, λύσεις για την αντιμετώπιση του σε επίπεδο Ευρωζώνης, γνωρίζετε το πρόταση για το Ταμείο Απόσβεσης του Χρέους. Ε, εσείς ως Προεδρεύον το ΕΚΟΦΗΝ, ε, στην προσπάθεια αυτή που κάνει η Ευρώπη για ανάκαμψη και τη διαφαινόμενη ανάκαμψη που έρχεται, ε, έχετε κάποιες προτάσεις κατά νου για την αντιμετώπιση του χρέους σε επίπεδο ευρωπαϊκό που φυσικά ε, θα έχει κάποιες ιδιαίτερες στοχευμένες ενέργειες για χώρες όπως είναι η δική μας η Ελλάδα. Αλλά επαναλαμβάνω είναι ένα ευρωπαϊκό πρόβλημα το δημόσιο χρέος και μάλιστα και στο, G20 στο οποίο θα συμμετέχετε ως Προεδρία και εκεί πιστεύω ότι είναι ένα θέμα το οποίο μπορείτε να θίξετε για αν θέλουμε να λέμε ότι είναι ειλικρινής η προσπάθεια της διεθνούς κοινότητας για ισορροπημένη ανάπτυξη και σταθερότητα στον κόσμο. Ευχαριστώ πολύ. Uh, Ευχαριστώ πολύ, Ρόδη. Ο τελευταίος ομιλητής είναι ο κύριος Γιώργος Τούσας. Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι, παρακολουθώντας ε, τις δύο μέρες της ε, διακυβερνητικής συνδιάσκεψης και σήμερα την ομιλία του κυρίου Υπουργού, του κυρίου Οικονομικών της Ελλάδας που έχει και την Προεδρία του ΕΚΟΦΗΝ ε, θέλω να επισημάνω ότι γίνεται μια έντονη προσπάθεια να προσδοθεί σε αυτή την διακυβερνητική διάσκεψη η δημοκρατική νομιμότητα των πολιτικών αποφάσεων που πάρθηκαν τα τελευταία 4,5 χρόνια στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διαφωνούμε πέρα ως πέρα και αποδεικνύεται από την ίδια την κατάσταση που επικρατεί στα 28 κράτη-μέλη η πλήρης αναντιστοιχία που υπάρχει μεταξύ αυτού που εκφράζεται εδώ στη συνεδρίαση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και από τους εκπροσώπους των ελληνικών κοινοβουλίων με την κατάσταση που ζουν 26 εκατομμύρια 700.000 άνεργοι 120 εκατομμύρια που ζουν κάτω από το όριο της στόχας στην πρώτη γραμμή νέοι από τις εργατικές λαϊκές οικογένειες. Ας είναι σίγουρο, με τεγνάσματα δεν πρόκειται να νομιμοποιηθεί στη συνειδήση των εργαζομένων αυτή η αντιλαϊκή πολιτική που την αντιπαλεύουν με όρους κινήματος και σε πολιτικό επίπεδο. Το δεύτερο στοιχείο που θα ήθελα να επισημάνω είναι το εξής. Ανάπτυξη. Για ποιον και με ποιο σκοπό. Είναι προφανής ότι η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ευρώπη 2020 έχει ως αφετηρία και κριτήριο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της κερδοφορίας των μονοπωλίων μέσα από την δραστική παραπεραμείωση της τιμής της εργατικής δύναμης. Δηλαδή το σύμφωνο για το ευρώ Plus θα χρησιμοποιηθεί μόνο για τους Έλληνες, τους Πορτογάλους, τους Ιρλανδούς και όποιους άλλους μπαίνουν σε συνθήκες επιτήρησης, οικονομικής επιτήρησης, μεσοπρόθεσης ή μακροοικονομικής επιτήρησης ή για το σύνολο των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μα είναι προφανές. Δεν μεταφράζω τη συνθήκη του Europlus. Κριτήριο σε ό,τι αφορά τις αμοιβέ των εργαζομένων πάβει να είναι οι συλλογικές συμβάσεις, τελειώνω κύριε Πρόεδρε, οι καδικές συμβάσεις εργασίας, οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας, αλλά η μονάδα κόστους εργασίας αναμονάδα παραγωγής του προϊόντος σε συγκεκριμένο χρόνο. Ισοπαίδωση των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης. Και τέλος είναι ένα ζήτημα ότι αυτή η εμβάθυνση της ΩΝΕ που χαρακτηρίζεται ε, και η Τραπεζιτική Ένωση κατά την άποψή μας θα ενισχύσει τις συγκέντρωση και συγκεντροποίηση του κεφαλαίου στο χρηματοπιστωτικό σύστημα και θα οξυθούν ακόμα παραπέρα οι αντιθέσεις τόσο μεταξύ των κρατών αλλά και των περιοχών. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα τώρα να ζητήσω από τους ομιλητές ακροατές που βρίσκονται, που κάθονται εδώ να θέσουν ερωτήσεις να ρωτήσω αν έχουν ερωτήσεις να θέσουν. Κυρία Περβάνος Περέζ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα τελειώνοντας να πω κάτι που αφορά τον θεμισμικό σκέλος του όλου θέματος. Εσείς θα πρέπει να φτάσετε στα υπόλοιπα συμπεράσματα. Θα ήθελα να αναφερθώ σε κάτι το οποίο μας απασχόλησε πάρα πολύ όλους σήμερα το πρωί και το οποίο δεν υπενθυμίστηκε εδώ στην Ολομέλεια σήμερα. Πριν από τις ε, ευρωεκλογές, στο κλίμα αυτό το οποίο ζούμε, πολλοί φοβούνται τον λανθάνοντα ευρωσκεπτικισμό, δεδομένου ότι πάρα πολλοί πολίτες ε, τους έχει καταστήσει αυτή η κρίση ιδιαίτερα ευάλωτους. Οι προσδοκίες λοιπόν των πολιτών μας είναι να τους δώσουμε σαφή μηνύματα για το ότι κατανοούμε τα προβλήματά τους για την ε, κοινωνική διάσταση του προβλήματος, για το ότι θα μπορέσουμε να θεσπίσουμε πραγματικά αυτή την εγγύηση για τους νέους και θα κάνουμε κάτι για την οικονομική ανάπτυξη. Αυτά ξέχασα να τα αναφέρω προηγουμένως, αλλά νομίζω όμως ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό το μήνυμα αυτό για τους συναδέλφους μετά από τις καρποφόρες αυτές συναντήσεις που είχαμε κατά τη διάρκεια των τρίων τελευταίων ημερών. Σας ευχαριστώ που με επιτρέψετε να κάνω αυτή την επισήμανση. Ευχαριστούμε πολύ και τέλος ο Πρόεδρος, ο Προεδρεύων του ΕΚΟΦΗΝ έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Στο ερώτημα του κυρίου Κρεμαστινού, ε, δεν ε, πιστεύω ότι υπάρχει ασυνέπεια μεταξύ αυτών που είπατε εσείς και, που, αυτών που είπατε ότι είπε ο κύριος Ολιρέν το να εγγυηθούμε φυσικά το 100.000 είναι όριο για όλους και για τον Βορρά και για τον Νότο ε, η, πρόθεση η πρόθεση αυτού του συστήματος είναι να προστατεύσει τους καταθέτες απόλυτα ε, διότι έχουμε, από την κρίση έχουμε μάθει, έχουμε πάρει αρκετά μαθήματα και δεν υπάρχει καμία διαφοροποίηση μεταξύ βορρά και νότου όσον αφορά το κομμάτι αυτό. Μιλάμε για προστασία όλων των καταθετών, είτε είναι στο βορρά είτε είναι στον νότο. Δεν υπάρχει απολύτως καμία διαφορά και η, εξασφάλιση της ομαλής ροής δανείων ε, προς επιχειρήσεις ακριβώς προϋποθέτει εμπιστοσύνη, γι' αυτό ακριβώς προωθούμε την Τραπεζική Ένωση ε, σε όλη την Ευρώπη. Όχι μόνο στο Βορρά, όχι μόνο στο Νότο, αλλά σε όλη, σε όλη την Ευρώπη. Ε, now on, the question raised by, Mr. Marini. Τώρα για το ερώτημα που έθεσε ο κύριος Μαρινή, σας διαβεβαιώ ότι η ελληνική προεδρία θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να ενισχυθεί ο διάλογος μεταξύ Προεδρίας και Εθνικών Κοινοβουλίων και Εθνικού Κοινοβουλίου και Ευρωπαϊκού με συγχωρείτε, Κοινοβουλίου για όλα τα θέματα ε, οικονομικής πολιτικής. Για αυτά που είπε η κυρία Τίσεν Ξέρουμε πολύ καλά ότι το Κοινοβούλιο δεν χαίρεται ιδιαίτερα σχετικά με... δεν είναι ικανοποιημένο με τη διακυβερνητική συμφωνία. Αλλά εδώ θα ήθελα να πω το εξής. αν συζητήσεις εδώ και πολλούς μήνες ε, οι οποίες τελικά οδήγησαν συμπεράσματα ε, κατά τα οποία αναλάβαμε τον ελάχιστο δυνατό κίνδυνο ή ρίσκο. Τι θέλουμε. Θέλουμε μια τραπεζική ένωση, ένα κεντρικοποιημένο σύστημα, έναν μηχανισμό εποπτείας και ένα μηχανισμό εξυγένσης. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα εμπλακεί σε κάθε στάδιο της δημιουργίας μιας ισχυρής τραπεζικής ένωσης. Εστε βέβαια. Now regarding Mr. Τώρα, το κύριο Σίλκιν έθεσε πολλά ερωτήματα για το ευρωπαϊκό εξάμεινο Βεβαίως, από τη μια υπάρχουν τα θέματα της σταθεροποίησης, δημοσιονομικής κτλ, απασχόλησης, κοινωνικής ε, συνοχής, η κατάσταση διαβελτιώθηκε τα τελευταία χρόνια. Εμείς τώρα θέλουμε να ε, δώσουμε έμφαση στις επενδύσεις, στη δημοσιονομική εξυγίανση που όμως να ενισχύει και τις πιθανότητες ανάπτυξης και να προσπαθήσουμε να εμπλέξουμε τους κοινωνικούς εταίρους στο διάλογο το σχετικό που θα γίνει. Και ναι βεβαίως ο στόχος της Τραπεζικής Ένωσης είναι να αποφύγουμε καινούργια κρίση των τραπεζών διότι όπως ξέρετε η κρίση της Ευρωζώνης εμπολίστανε κρίση των τραπεζών. Πρέπει να προσέξουμε πολύ βεβαίως για να δούμε από τη μια για να είμαστε εξισορροπημένοι στην προσέγγιση μας Ως Έλληνας Υπουργό Οικονομικών και όχι ως ε, Πρόεδρος του ΕΚΟΦΗΝ εδώ, γιατί αφορά την Ελλάδα. Ε, ε, έχω την την, απάντηση του κυρίου Ντάιζεμπλουμ στο Ολλανδικό Κοινοβούλιο. Αναγνωρίζει ότι υπάρχει πολύ μεγάλη πρόοδο αν διαβάσετε την απάντησή του, ε, ότι όσον αφορά την εκταμείωση των προαπαιτημένων ε, είχαν τηρηθεί όλα τα προαπαιτούμενα του, του Δεκεμβρίου, αλλά βεβαίω αναφέρει ότι υπάρχουν ακόμα μερικέ εκκρεμότητε. Αυτέ τι εκκρεμότητε ε, κουβεντιάζουμε τώρα με την ε, Τρόικα. Ε, καθώς βρισκόμαστε προ το τέλο του, του προγράμματος, αυτό είναι ένα δύσκολο review. Ε, Προσπαθούμε λοιπόν ε, ως ελληνική κυβέρνηση ε, να πετύχουμε το καλύτερο δυνατό για τον ελληνικό λαό. Γι' αυτό οι διαπραγματεύσεις αυτές ε, με την Τρόικα θα κρατήσουν όσο πρέπει να κρατήσουν, αλλά μην ανησυχείτε, στο τέλος όπως έχει γίνει μέχρι σήμερα θα έχουμε, θα έχουμε συμφωνία. Τώρα, ε, όσον αφορά την ε, Τρόικα, οι, οι, οι θέσεις της ελληνικής κυβέρνησης έχουν αποτυπωθεί στην απάντηση που έστειλα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με πολύ μεγάλη λεπτομέρεια. Ε, νομίζω είναι, είναι δημοσιευμένη, είναι και στο site και του, και του Ελληνικού Κοινοβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου οι απόψεις μου και οι απόψεις της ελληνικής κυβέρνησης είναι εκφρασμένες εκεί. Θέλω να πω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λογοδοτεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με τις ε, δραστηριότητες της Τρόικας ε, στις χώρες μέλη. Ε, είμαστε ανοιχτοί σε προτάσεις, σε διαδικασίες, πάντοτε όσον αφορά την δημοκρατική νομιμότητα και τη δημοκρατική νομιμοποίηση. Όσον αφορά το χρέος, και αυτό το ερώτημα επίσης έκανε και η κυρία Ρόδη Κράτσα και ο κύριος Τούσας, κατά την άποψή μου, επειδή ρωτήσατε την, άποψή μου, ο πιο ασφαλής τρόπος για να μειωθεί ο λόγος του χρέους είναι να επιτύχουμε και πάλι στην Ευρώπη υψηλούς ρυθμούς οικονομικής ανάπτυξης. Ε, αυτό είναι το υπαριθμόν ένα για μένα, ο ε, υπαριθμόν ένα τρόπος ε, για να μειωθεί το, το χρέος και ο, και ο πλέον βιώσιμος τρόπος. φυσικά υπάρχουν και, άλλες, υπάρχουν και άλλοι, και άλλοι, και άλλοι, και άλλοι τρόποι. Η ιδιωτικοποίηση για παράδειγμα είναι ένας, είναι ένας τρόπος. Ε, όπου εκεί πέρα πετυχαίνει και μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα ε, και έσοδα για την ε, μείωση του χρέους. Τώρα, όσον αφορά την Ελλάδα, αφορά το ερώτημα της κυρίας, της κυρίας Κράτσα, όπως ξέρετε στο Eurogroup του Νοεμβρίου του 2012 υπάρχει μια νομική βάση για περαιτέρω μείωση του, του χρέους με τους κατάλληλους τρόπους ε, εφόσον τηρηθούν ορισμένες προϋποθέσεις και η βασικότερη προϋπόθεση είναι ε, να πετύχει η Ελλάδα πρωτογενές πλεόνασμα. Η Ελλάδα πέτυχε πρωτογενές πλεόνασμα το 2013. Περιμένουμε λοιπόν τώρα να τελειώσουμε ε, την επισκόπηση που κάνει η Τρόικα, ούτω ώστε στο Eurogroup να ξεκινήσουμε και τη συζήτηση αυτή για τη βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους σχετικά με τα άλλα ερωτήματα που έθεσε η κυρία Κράτσα, πράγματι πρέπει να κοιτάξουμε τη χρηματοδότηση της οικονομίας. Όπως είπα στην ομιλία μου, εκεί δεν είχαμε δώσει αρκετή έμφαση σε προβλήματα ρευστότητας. Πολλά οικονομικά μοντέλα που είχαν χρησιμοποιηθεί δεν είχαν λάβει υπόψη αυτή την παράμετρο. Τώρα έχουμε γίνει σοφότεροι από την κρίση, βέβαια με τη σοφία της ύστερης γνώσης και καταλαβαίνουμε την πολύ μεγάλη σημασία που έχει χρηματοδότηση, εξού και βασική έμφαση ε, δίνεται στην Τραπεζική Ένωση. Ε, εξού και βασική έμφαση δίνεται στο ρόλο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, του, του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων, στο να εξασφαλίσουμε αρκετά κεφάλαια για την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων που θα, που θα πρέπει να διοχετευθούν κυρίως σε περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν πρόβλημα, που έχουν πρόβλημα ανεργίας, που έχουν πρόβλημα χαμηλής οικονομικής ανάπτυξης, αλλά και που δίνουν ευκαιρίες. Ε, Η απάντησή μου στον κύριο Παπαδημούλη ως προς το χρέος αφορά και την Ευρώπη και την Ελλάδα κατά τον ε, ειδικότερο τρόπο. Ε, τέλος, ε, στα ερωτήματα που έθεσε ο κύριος ε, ε Τούσιας, εγώ πιστεύω κύριε Τούσια ότι η εμπάθηση της ΟΝΕ θα ωφελήσει τον πολύ κόσμο. Δεν είναι, δεν είναι μια πολιτική η οποία θα θα ωφελήσει το κεφάλαιο σε βάρος εργαζομένων. Πιστεύω ότι με την, ε, εμβάθυνση της ΟΝΕ, ε, με μια αποτελεσματικότερη τραπεζική ένωση, ε, με, μια, με έναν συντονισμό των οικονομικών πολιτικών θα έχουμε και μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και μεγαλύτερη κοινωνική δικαιοσύνη. Δέστε στο, στο ευρωπαϊκό ε, εξάμεινο τώρα ακριβώς πόσο πιο ισορροπημένη είναι η προσέγγιση μεταξύ δημοσιονομικής προσαρμογής, ε, μεταξύ δημιουργίας θέσεων εργασίας και τέλος ε, κοινωνικής συνοχής. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ τον Έλληνα Υπουργό των Οικονομικών και Πρόεδρο του ΕΚΟΦΗΝ και τώρα δίνω το λόγο στον Αντιπρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τον κύριο Κάρας. Αγαπητέ συνάδελφε Τραγάκη, κύριε Υπουργέ, αξιότιμες κυρίες και κύριοι, θα ήθελα στο τέλος αυτής της τριήμερης διάσκεψης να ευχαριστήσω όλους τους ευρωβουλευτές άσχετα από το ποια χώρα προέρχονται, από ποιο κοινοβούλιο προέρχονται για την ενεργή συμμετοχή τους και την παρουσία τους. Αυτό που βιώσαμε εδώ τις τελευταίες τρεις μέρες δεν είναι τέλειο αλλά σίγουρα είναι ένα βήμα μπροστά. Είναι μια πρεμιέρα από πολλές ε, οπτικές γωνίες. Πρώτα-πρώτα, λαμβάνει χώρα μια συνδιάσκεψη όπου τα θέματα του άρθρου 13 του Δημοσιονομικού Συμφώνου συνδέονται με τη συζήτηση για το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Κοινοβουλευτικής Εβδομάδας. Μέχρι τώρα είχαμε κάνει εκδηλώσεις στο Βίλνιος ας πούμε για το άρθρο 13 ή πέρσι εδώ στο Κοινοβούλιο για το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο. Τούτη τη φορά όμως, για πρώτη φορά και τα δύο αυτά συνδέονται και οι δύο αυτές συζητήσεις γίνονται παράλληλα και από κοινού. Ίσως ορισμένοι πιστεύουν ότι είναι υπερβολικό αυτό. Άλλοι ίσως πιστεύουν ότι αυτό δεν αρκεί. Ωστόσο βλέπουμε ότι η συζήτηση για το Δημοσιονομικό Σύμφωνο το θέμα του δημόσιου χρέους και η μείωση του δημόσιου χρέους συνδέονται στενότατα με τα γενικά κότερα ζητήματα με τη δημοσιονομική πολιτική, τα προγράμματα απασχόλησης κτλ. Με άλλα λόγια, με την πολιτική μας ευθύνη έναντι της κοινωνίας. Είναι καλό αυτό κατά την άποψή μου, γιατί καταφέραμε μαζί να συνδέσουμε το δημοσιονομικό σύμφωνο με το ευρωπαϊκό εξάμεινο και να τα κουβεντιάσουμε μαζί. Δεύτερο, για πρώτη φορά η συνδιάσκεψη αυτή έχει διάρκεια τριών ημερών. Και από ό,τι γνωρίζω η συμμετοχή ήταν τεράστια, πολύ μεγάλη. Δεν ξέρω, μπορεί κάποιοι να έλειπαν γιατί είχαν αλλημένες υποχρεώσεις, αλλά η παρουσία όλων αυτών των ανθρώπων αυτές τις μέρες δείχνει και στην κοινή γνώμη ότι οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι των ευρωπαϊκών λαών αγωνίζονται για την εντατικοποίηση του διαλόγου και παίρνουν πολύ σοβαρά τα θέματα τα οποία ανησυχούν τον πολίτη. Αυτό είναι η δουλειά μας τελικά. Τρίτο θέμα, κάποιος είπε κάτι τι και με ενόχλησε λίγο Κανείς μας δεν ελέγχει τον διπλανό του. Όλοι ελέγχουμε τις κυβερνήσεις. Ό,τι κάναμε το κάναμε μαζί. Δεν νομίζω ότι η ελληνική προεδρία έχει την αίσθηση ότι ελέγχεται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ούτε εμεί, κανείς έχει την αίσθηση ότι η Ελληνική Προεδρία ελέγχει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Από κοινού δουλεύουμε, δουλεύουμε μαζί για να προχωρήσουν ορισμένα θέματα. Και σας ευχαριστώ γι' αυτό. Και το άλλο σημαντικό που πρέπει να έχουμε στο νου μας είναι ότι όλα εδώ συμβαίνουν μέσω συμβιβασμών. Αλλά καμιά φορά δεν χρειάζεται συμβιβασμός. Γιατί ε, όταν γνωρίζουμε καλά την Ευρωπαϊκή Ένωση, όταν οι στόχοι είναι... Ε, ε, στόχοι τους οποίους υποστηρίζουν όλοι. Και εδώ εμείς απλώς κάνουμε τη δουλειά συντονιστή, δεν χρειάζεται συμβιβασμοί. Έχουμε εκατοντάδες εκπροσώπους εδώ των διαφόρων κοινοβουλίων, των διαφόρων χωρών μελών και η πείρα μας δείχνει ότι έχουμε ε, πολλά να μάθουμε ένας από τον άλλον. Χτες παραδείγματος χάρη ήρθε η εκπρόσωπος του Ισδανικής Βουλής του Φολκετινγκ στο γραφείο μου και μου είπε ότι αυτό το οποίο ονομάζουμε εμείς Ευρωπαϊκή Εβδομάδα θα το, επαναλα... θα το μιμηθεί το Ευρωπαϊκό το Δανικό Κοινοβούλιο και θα ξεκινήσει μια Δανέζικη Κοινοβουλευτική ε, εβδομάδα. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό και θα κάνει ένα δανεικό εξάμεινο. Πώς μπορεί να μετατραπεί λοιπόν το ευρωπαϊκό εξάμεινο σε εθνικά εξάμεινα. Αυτό είναι μια πολύ καλή ιδέα. Γνωρίζουμε πολύ καλά όλοι μας ότι αυτούς τους κοινού ε, στόχους μπορούμε να τους επιτύχουμε μόνο εάν εφαρμόσουμε τις ε, ε, ειδικές αναχώρες και ε, αλλά θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι για το έτος 2012 μόνο 15% των συστάσεων αυτών ε, εφαρμόστηκαν. αν δεν δημιουργήσουμε λοιπόν τις περιστάσεις και τους όρους που να μας οδηγήσουν στο να μπορέσουμε να ε, εφαρμόσουμε το σύνολο των συστάσεων ποτέ δεν θα ε, επιτύχουμε τους κοινούς στόχους. Και εδώ θα ήθελα να πω ότι ε, να ε, συζητήσαμε ε, για το ρόλο των κοινοβουλίων ε, που δεν είναι λόγο μιλάμε για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εναντίον των Εθνικών για τα Εθνικά εναντίον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εμείς είμαστε οι εκπρόσωποι των πολιτών της Ευρώπης δεν υπάρχει ή το ένα ή το άλλο κοινοβούλιο είμαστε όλοι εκπρόσωποι των πολιτών μας και γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό η αρχή της συνένεσης να είναι το κύριο χαρακτηριστικό των εργασιών μας και όχι η αντιπαράθεση των μεν με τους δε. Έχουμε μια κάποια ευθύνη έναντι στους πολίτες μας, έναντι στις κυβερνήσεις, έναντι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα πρέπει να δουλέψουμε όλοι μαζί Γι' αυτό ευχαριστώ για άλλη μια φορά για τη δουλειά που έγινε αυτές τις τρεις μέρες όπου δουλέψαμε όλοι μαζί. Εκείνο που είναι σημαντικό είναι να μην τσακωνόμαστε ο ένας με τον άλλο, να μην φοβόμαστε ο ένας με τον άλλο, να επιτύχουμε κοινού στόχους, στόχους που κουβεντιάσαμε όλοι μαζί. Κυρίες και κύριοι, δεν είναι σωστό ότι η έκθεση Λικάνεν <laughs> μπήκε στο σιρτάρι. Το θέματα της έκθεσης Λικάνεν τελικά ε, ε, θα πρέπει να τα χρησιμοποιήσουμε, τα συστήσουμε, να τα εφαρμόσουμε ίσως. Να βοηθήσει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τίποτα δεν μπήκε στο σιρτάρι ή στον κάλαθο των αχρήστων. Και είναι γεγονός. Μιλάμε για τραπεζική ένωση. Ε, γιατί για να αποφύγουμε την επόμενη κρίση τραπεζών. Λοιπόν, θα μπορούσαμε να κάνουμε μια δημοσιονομική, μια ένωση των προϋπολογισμών, δημοσιονομική ένωση για να αποφύγουμε αντίστοιχη κρίση στο μέλλον. Όλοι μαζί μπορούμε να προχωρήσουμε και αυτή η αίθουσα το δείχνει αυτό το δείχνουν οι τελευταίες τρεις μέρες ας συνεχίσουμε να οδεύουμε μαζί στην ίδια πορεία και να προσπαθούσουμε όλοι μαζί να σαν Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σαν καρδιά της Ευρωπαϊκής Δημοκρατίας να βοηθήσουμε βοηθήσουμε τους πολίτες μας. Auf Wiedersehen στη Ρώμη. Last but not least. Και τέλος, νομίζω ότι θα πρέπει να δώσουμε το λόγο στον κύριο Τραγάκη. Κύριε Αντιπρόεδρε, η διακοινοβουλευτική διάσκεψη για την οικονομική διακυβέρνηση ευρωπαϊκής ένωσης στα πλαίσια της ευρωπαϊκής εβδομάδας νομίζω κατά τη γνώμη μου ότι εστέφθη από απόλυτη επιτυχία. μέρος της επιτυχίας αυτής πιστώνεται και σε εσάς κύριε αντιπρόεδρε κύριε κάρας. συμμετείχαν περίπου 150 βουλευτές εθνικών κοινοβουλίων ή ευρωβουλευτές και είχαμε 30 ομιλητές και περίπου 100 παρεμβάσεις. Στο τριήμερο αυτό είχαμε την ευκαιρία να ανταλλάξουμε απόψεις πάνω σε θέματα πρώτης γραμμής σχετικά με την οικονομική διακυβέρνηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωζώνη. Μιλήσαμε για την εμβάθυνση της ΟΝΕ και την Τραπεζική Ένωση, στην οποία κυρίως επισπεύδεται η συζήτηση στην περίοδο αυτή και με την οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει την ευκαιρία να διορθώσει λάθη και παραλήψεις των τελευταίων ετών με την επαναξιολόγηση της υφιστάμενης δομής και κινήτρου λειτουργίας του ευρωπαϊκού τραπεζικού τομέα. Οι ευθύνε για μεταρρυθμίσεις που έχουν ως στόχο την αποτελεσματικότερη εποπτεία και εξυγίανση των πιστοτικών ιδρυμάτων είναι μεγάλες. Παράλληλα όμως οι ευκαιρίες για την επίτευξη μιας αποτελεσματικής τραπεζικής ένωσης προς όφελος του κοινωνικού συνόλου είναι ακόμα μεγαλύτερες. Η πλήρης τραπεζική ένωση είναι φυσικά αναγκαία, αλλά όχι επαρκής. Απαιτείται επιπλέον η δημοσιονομική και οικονομική ενοποίηση και τέλος η πολιτική μέσω έντονης συνεχούς διαβούλευσης μεταξύ θεσμικών φορέων που θα ενισχύσει τη δημοκρατική νομιμότητα όλων των αποφάσεων που λαμβάνονται σε κεντρικό επίπεδο. Σε αυτή την κατεύθυνση εξέχοντα ρόλο θα πρέπει να διαδραματίσουν τα κοινοβούλια μας σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η κοινωνική διάσταση από την άλλη θα πρέπει να αποτελεί αναπόσπαστο μέλος αυτής της διαδικασίας ούτως ώστε να αποδείξουμε στους πολίτες που εκπροσωπούμε ότι λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη τις κοινωνικές συνέπειες που δημιουργούν οι περιοριστικές πολιτικές που ακολουθούμε σε πολλές χώρες Ευρώπης. Η επιτυχής έκβαση αυτής της προσπάθειας θα θέσει οριστικό τέλος στην αστάθεια και την αβεβαιότητα που παρατηρείται ιδίως σε χώρες περιφέρειας. Ο παναπροσδιορισμός του τρόπου με τον οποίο οι ευρωπαϊκές τράπεζες στηρίζουν την πραγματική οικονομία μπορεί να επιτευχθεί με την εφαρμογή κατάλληλων ρυθμίσεων διασφαλίζοντας παράλληλα τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα για τη στήριξη της πραγματικής οικονομίας κομβικής σημασίας είναι επίσης η εφαρμογή του συμφώνου ανάπτυξης για την απασχόληση όπως και ειδικέ δράσεις κατά πολέμης ανεργίας ιδίως των νέων που έχουν φτάσει σε πρωτόγνωρα υψηλά επίπεδα και την προώθηση των επενδύσεων σε κέρους τομείς όπως παραδείγματος χάρη τα μέτρα που αποφασίστηκαν στο Συμβούλιο του Ιουνίου για τους ανέργους και το επενδυτικό σχέδιο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και της Επιτροπής για τη Χρηματοδότηση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων της Περιφέρειας. Η μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας μέσω εναλλακτικών πηγών πέραν του στενού χρηματοπιστωτικού συστήματος εξετάζεται τον τελευταίο καιρό και είναι αυτό ένα ακόμη θετικό βήμα. Η δομική και άρρηκτη σχέση ανάπτυξης και απασχόλησης πρέπει πάντοτε να λαμβάνεται υπόψη για την επίτευξη της κοινωνικής και οικονομικής συνοχής των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο κίνδυνος μιας άνεργης ανάπτυξης πρέπει πάση θυσία να εξαλειφθεί και έτσι χρειάζεται να εφαρμόζεται το κατάλληλο μείγμα πολιτικών δημοσιονομικής σταθερότητας και πολιτικών φιλικών προς την ανάπτυξη που θα διέπεται από την κατάλληλη ευελιξία και θα αναπροσαρμόζεται ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούν. Χθες εξετάσαμε επίσης τη δημοκρατική νομιμότητα των προγραμμάτων οικονομικής προσαρμογής. Στις περιόδους οικονομικής λιτότητας που διανύουμε είναι πολύ σημαντικό να φαίνεται ξεκάθαρα η αναγκαιότητα και οι προοπτικές αλλά και η αποτελεσματικότητα των μέτρων που λαμβάνονται στα πλαίσια της δημοσιονομικής εξυγείας. Έτσι μόνο οι πολίτες θα μπορέσουν να δεχτούν την όποια μείωση του βιωτικού τους επίπεδου και να υποστούν θυσίες. Πρέπει κατά το σχεδιασμό των σχετικών μέτρων να υπάρχει διάλογος με όλους τους αρμόδιους κοινωνικούς φορείς και τα θεσμικά όργανα. Η μέχρι τώρα πορεία εφαρμογής και η εμπειρία μας εφαρμογής των προγραμμάτων δημοσιονομικής προσαρμογής έχει δείξει ότι τα μέτρα που έχουν πάρθει έχουν άμεσο αρνητικό αντίκτυπο στην απασχόληση και την κοινωνική συνοχή. Οι πολιτικές αυτές αυστηρής λιτότητας που επιβάλλουν τα εν λόγω προγράμματα πρέπει να καθοδηγούνται από τις συνθήκες της Ένωσης που επιτάσσουν προώθηση της απασχόλησης, προώθηση της εκπαίδευσης και υγείας και της απαραίτητης κοινωνικής προστασίας αλλά και να συμπλέουν με τις προτεραιότητες της στρατηγικής 2020. Τα εθνικά κοινοβούλια και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με τους άμεσα εκλεγμένους αντιπροσώπους τους. Πρέπει να κατέχουν ενεργό ρόλο στις διαβουλεύσεις με την Τρόικα. Πριν την επιβολή των προγραμμάτων αυτών και να εφαρμόζονται πιστά οι νόμιμες διαδικασίες μέχρι τη στιγμή της ψήφισης των προγραμμάτων από τα κοινοβουλευτικά σώματα. Η διαδικασία του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου μπορεί να έχει ξεκινήσει από το 2011 αλλά χρόνο με το χρόνο ότι αντιμετωπίζονται αρκετές ανεπάρκειες και ότι υλοποιούνται απαραίτητες συμπληρωματικές ενέργειες. Οι ξεκάθαρα ειδικά προσαρμοσμένες για κάθε χώρα συστάσεις με ποιοτικούς και ποσοτικούς στόχους αφήνοντας πάντα ευελιξία κινήσεων στα κράτη-μέλη αποτελούν μια σημαντική θετική εξέλιξη. Η παρακολούθηση των συστάσεων και ο έλεγχος εφαρμογής που έλειπε από τους προηγούμενους κύκλους των ευρωπαϊκών εξαμήνων που εφαρμόστηκε για πρώτη φορά τον περασμένο Οκτώβριο φαίνεται ότι επέφερε τα επιθυμητά αποτελέσματα μιας και όλα σχεδόν τα κράτη-μέλη αλλά περισσότερο και άλλα λιγότερο εμφανίστηκαν συμμορφωμένα προς τις συστάσεις που είχαν εκδοθεί αναπερίπτωση. Κατά το τρέχον ευρωπαϊκό εξάμεινο θα χρησιμοποιηθούν για πρώτη φορά κοινωνικοί και εργασιακοί δείκτες σε σχέση με την κοινωνική διάσταση της Ευρωζώνης και θα υπάρξει στενότερη συνεργασία με των Εθνικών Κοινοβουλίων και της Επιτροπής πριν από το δημοσίευση των αναχώρα συστάσεων. Ιδιότερη προσοχή πρέπει να δοθεί και στα μακροχρόνια διαρθρωτικά προβλήματα που επηρεάζουν την μακροοικονομική θέση των κρατών μελών και την ανταγωνιστικότητά τους και καταδεικνύονται μέσω της διαδικασίας μακροοικονομικών ανισορροπιών που συμπληρώνει τη διαδικασία του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Τα τελευταία χρόνια έχουν σημειωθεί αποκλίνουσες οικονομικές τάσεις που δημιούργησαν χάσμα ανταγωνιστικότητος μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που όμως το τελευταίο έτος έχουν ξεκινήσει να εξομαλύνονται. Είναι θετική η πρόταση της Επιτροπής για συμπερίληψη βασικά πίνακα βασικών κοινωνικών και εργασιακών δικτών στη διαδικασία. Πρέπει όμως οι δείκτες αυτοί να αντικατοπτρίζουν επαρκώς την πραγματική εικόνα των κρατών μελών σε αυτούς τους τομείς αλλά και τη μεταξύ τους αλληλεξάρτηση. Η αντιμετώπιση των ανισορροπιών είναι κλειδί για τη σταδιακή ανάκαμψη και σύγκληση των ευρωπαϊκών οικονομιών. Ιδιαίτερα ενδιαφέρον είχαν και τα συμπεράσματα από τις σημερινές συνεδριάσεις των τριών επιτροπών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Για να συνοψίσω, ως βασική τομής προτεραιότητας για τη μελλοντική οικονομική διακυβέρνηση θα πρέπει να είναι πρώτον μείγμα πολιτικών που θα προωθούν την ανάπτυξη ιδίως για τις χώρες που βρίσκονται σε ύφεση και το οποίο δεν θα θέτει σε κίνδυνο τη δημοσιονομική εξυγίανση αλλά θα ενισχύει την ανταγωνιστικότητα, την απασχόληση και τις επενδύσεις. Δεύτερον, ενοποιημένο δημοσιονομικό πλαίσιο που θα διασφαλίζει τη χάραξη ορθής δημοσιονομικής πολιτικής σε εθνικό αλλά και ευρωπαϊκό επίπεδο βάσει συντονισμού και κοινή λήψη αποφάσεων. Τρίτον, ενοποιημένο χρηματοοικονομικό πλαίσιο που περιλαμβάνει εποπτεία σε ευρωπαϊκό επίπεδο και κοινού μηχανισμούς εξυγίανσης των τραπεζών και εγγύηση των καταθέσεων για τη διασφάλιση οικονομικής σταθερότητας και ελαχιστοποίηση του κόστους αποτυχίας των τραπεζών στις πλάτες των φορολογούμενων πολιτών. Κοινή πολιτική στήριξη της ρευστότητας των αγορών, ιδίως για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας είναι πολύ σημαντικός σε αυτό το πλαίσιο. Τέλος, διασφάλιση της απαραίτητης δημοκρατικής νομιμότητας και λογοδοσίας των αποφάσεων που λαμβάνονται σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα βασίζεται στην κοινή άσκηση κυριαρχίας για κοινέ πολιτικές και στην αρχή της αλληλεγγύης. Κλείνοντας θα ήθελα να πω δύο λόγια για αυτή εδώ τη συνδιοργάνωση που αποτελεί ένα νέο παιδί της διακοινοβουλευτικής συνεργασίας πραγματοποιήθηκε μετά από πολύμηνη εντατική συνεργασία σε πολιτικό και διοικητικό επίπεδο με διαφωνίες και συμφωνίες προσπαθώντας να συγκεράσουμε την ευρωπαϊκή με την εθνική πολυπλοκότητα αλλά με έναν και μόνο γνώμονα τη συμπληρωματικότητα και την κοινή στόχευση των εθνικών κοινοβουλίων που δεν είναι άλλη από τη στήριξη της ενωμένης ευρωπαϊκής μας πορείας και των συμφέρων των πολιτών που όλοι εμείς εδώ εκπροσωπούμε. Αποφασιστικό ρόλο γι' αυτό έπαιξε και ο αντιπρόεδρος ο κύριος Κάρας με τον οποίο είχαμε πράγματι μια πολύμινη συνεργασία για αυτό το νέο πεδίο όπως το ονόμασα. Δεν βλέπω τον κύριο Μαρινή εδώ, αλλά ήθελα, ήθελα επειδή το, επέθε, το έθεσε ερώτηση, υπενθυμίσω, το ανάλυσα και χτες, το ανέλησα και χτες, το είπε και ο κύριος Κάρας, ότι θα ενημερωθείτε πιο αναλυτικά για τον οδικό χάρτη που από τον επόμενο μήνα θα επανεκκινήσει τις διαδικασίες σχετικά με τον κανονισμό λειτουργίας της διάσκεψης για την οικονομική διακυβέρνηση ένα κανονισμό που θα έχει σαν στόχο τη διασφάλιση της εύρυθμης και αποτελεσματικής λειτουργίας της διάσκεψης αυτής. Με αυτά τα λόγια θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αλλά και των Εθνικών Κοινοβουλίων και όλους εσάς για την παρουσία σας και όχι μόνο αλλά κυρίως για την ενεργό συμμετοχή σας. Σας ευχαριστώ πολύ.